Euh, Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Donc, je vous souhaite à tous euh, la bienvenue pour notre euh, réunion. Καλώς ήλθατε όλες και όλοι στη συνεδρίαση αυτή. Με μεγάλη σας ξαναβρίσκω μετά από μια μακρά απουσία. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που με αντικατέστησαν στην Προεδρία της Επιτροπής, ιδίως την κυρία Πφεφέ, την κυρία Κρετέλ, τον κύριο Ντέβα. Σας ευχαριστώ όλους. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν δύο αιτήσει για τροποποίηση της ημερήσιας αυτής διάταξης. Ο κύριος ε, Ζαχραντήλ, η ψηφοφορία για την άκτα θα αναβληθεί στις, μέχρι τις 4 Ιουνίου, κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα γιατί η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Ίντα ψηφίζει στις 20 Ιουνίου. Επίσης, αιτήσει του εισηγητού κυρίου Πόγκα θα προτείνω να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξή μας την ψηφοφορία της έκθεσής του για την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με την τροποποίηση της απόφασης 2001 κάθετος 822 του Συμβουλίου σε σχέση με την Ένωση των χωρών και εδαφών, των υπερπόντιων χωρών και εδαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια αλλαγή του ευρωπαϊκού καθεστώτος του Αγίου Βαρθολομέου του Σαν που έλαβε χώρα στην 1η Ιανουαρίου 2012 από υπερπεριφερική περιοχή σε χώρα και διαμέρισμα υπερποντίου χαρακτήρους. Οι σκιώδεις εισηγητές και οι πολιτικές ομάδες έχουν πληροφορηθεί με email για την αίτηση αυτή του κυρίου Πόγκα. Έχετε σχόλια ή αντιρρήσεις για την ημέρηση διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί, όχι, τότε εγκρίνεται. Και τώρα θα πάμε στα πρακτικά της συνεδρίασης 23 και 24 Απριλίου 2012 που έχουν διανεμηθεί στους φακέλους σας. Εάν έχετε σχόλια σε σχέση με αυτά τα πρακτικά, θα πρέπει να τις αναφέρετε στη γραμματεία μέχρι το τέλος της σημερινή μας συνεδρίασης. Αλλιώς θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Στη συνέχεια, έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών από την Δευτέρα Απριλίου 2012. Έχετε στο φάκελό σας τις συστάσεις αυτές και τις αποφάσεις της ηλιμένες των συντονιστών στις 24 Απριλίου 2012. Αν έχετε λοιπόν σχόλια σε σχέση με τα συμπεράσματα αυτής της συνεδρίας των συντονιστών, παρακαλώ να τα αναφέρετε στους, στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασης. Ο κύριος Φρανκ Φαν εκ έχει θέσει ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη χρηματοδότηση των εκλογών, την εν μέρη χρηματοδότηση των εκλογών στη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν τον βλέπω τον Φρανκ όμως στις τάξεις μας. Είναι η δεύτερη φορά που αποσιάζει όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στην Κομισιόν. Προτείνω να τεθεί αυτό το ερώτημα εγγράφως από τον κύριο Φανέκη από την Κομισιόν η οποία θα πρέπει να απαντήσει εγγράφως με αντίγραφο στη γραμματεία ώστε να διανύμουμε και εμείς τις απαντήσεις της Κομισιόν. Προχωρούμε τώρα στην εξέταση της τροποποίησης οδηγίας 2004 109 για την εναρμόνιση των υποχρεώσεων διαφάνειας σε σχέση με τις υποχρεώσεις των εκδοτών κινητών αξιών που οι κινητές αυτές αξίες είναι υποδιαπραγμάτευση σε, μια, ε, σε ένα χρηματιστήριο και τις οδηγίες 2007 καθώς 14 της Επιτροπής. Η συγγήτρια για τα θέματα αυτά είναι η κυρία Φιώνα Χολ της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Πρόκειται για την οδηγία λοιπόν για τη διαφάνεια και την ε, έκθεση για τις αιτήσει οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών. Και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος των εκθέσεων αυτών είναι να αυξήσουν τη διαφάνεια και να μειώσουν την φοροδιαφυγή. Εγώ σας προτείνω να τις συζητήσουμε από κοινού τις δύο εκθέσεις. Να τονίσω επίσης ότι αυτή είναι και αυτή η εργασία, αυτές οι δύο οδηγίες είναι απόρρια προσπαθειών πολλών ΜΚΟ και πολλών κοινοβουλευτικών. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά δίνω στην Φιώνα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και για την σύσταση το 5 και το 6 να τα δούμε μαζί. Νομίζω ότι είναι τελείως λογικό. Αυτό που αφορά ιδιαίτερα εμάς είναι το κεφάλαιο 9 της οδηγίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 και της οδηγίας διαφάνειας. Η νόμ είναι η αρμόδια επί της ουσίας και εμείς απλώς νομοδοτούμε μαζί με άλλες επιτροπές. Θα έχετε δει από το ηλεκτρονικό μήνυμα των, προς όλα τα μέλη μας ότι οι άλλες επιτροπές επιταχύνουν τη διαπαιρέωση για να τελειώσει η διαδικασία μέχρι το τέλος Ιουνίου, αν και δεν είναι βέβαιο αυτό. Σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και ότι η διορία κατάθεση των τροπολογιών θα λήξει αύριο το μεσημέρι, αν κατάλαβα καλά. Καταρχήν το ιστορικό. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου είναι ουσιώδης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα μπορούσαν να γεννήσουν δισεκατομμύρια σε φόρους. Αλλά επίσης οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν εκμεταλλεύονται όπως θα έπρεπε τις πηγές τους όπως η Νιγηρία που είναι πολύ πτωχότερες και ασταθέστερες από ό,τι θα μπορούσαν να είναι. Και δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για από τις κυβερνήσεις και τις εξορρυκτικές εταιρείες. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των εταιριών αυτών για να μπορέσουν οι πολίτες να ε, κρατούν την κυβέρνηση υπόλογη ως προς τη χρήση του ορυκτού της πλούτου. Οι χώρες που έχουν πολλούς πόρους αλλά δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη πρέπει να τύχουν μιας δίκαιας μεταχείρισης. Προς η ενωσιακή νομοθεσία δεν απαιτεί από τις εταιρείε αυτές να δίνουν αυτές τις πληροφορίες και να κάνουν τις πληρωμές τους σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια, αν και θα μπορούσαν να βελτιώσουν έτσι πάρα πολύ τους πόρους της χώρα, των χωρών αυτών. Από το 7 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει προτάσεις για αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών από τις εταιρείες αυτές το 11 η Κομισιόν υπέβαλε προτάσεις διόρθωσης της οδηγίας για τη διαφάνεια και ιδιαίτερα για τους λογαριασμούς των εταιρείων. Η προτινόμενη νομοθεσία απαιτεί από όλες τις εξορυκτικές εταιρείες που είναι γραμμένες στον επίσημο ενωσιακό κατάλογο καθώς και σε μη εγγεγραμμένες θα τις υποχρεώνει να δημοσιεύουν τους λογαριασμούς τους στις κυβερνήσεις για οποιαδήποτε εξορρυκτική ή δασοκομική δραστηριότητά τους σε όλες τους τις χώρες, σε όλες τις χώρες όπου δρούν. Αυτό θα έδινε στους πολίτες σε πλούσιες, σε πόρους χώρες αλλά υπανάπτυκτες περισσότερες πληροφορίες για καλύτερη διακυβέρνηση και λιγότερη διαφθορά αλλά επίσης θα ωφελούσε και τους επενδυτές και επενδύτριες που θα γνώριζαν έτσι καλύτερα την κατάσταση και τη λειτουργία των, χωρών, των εταιριών αυτών. Θα συμπλήρωνε δηλαδή αυτά που έχουμε ήδη προβλέψει για την πρωτοβουλία διαφάνειας των εθελοντικών λεγόμενων εξορρυκτικών εταιριών. Το 10, το νομοθέτημα Dodd-Frank απαιτεί από την Επιτροπή ομολο... Ομολόγων και Χρηματιστηρίου τέτοιες είδους αποκαλύψεις. Και οι προτάσεις της Κομισιόν είναι σωστές, αλλά κατά τη γνωμοδότησή μου προτείνω και μερικές αλλαγές σε ορισμένα σημεία για να υπάρξει κάποια βελτίωση. Ορίστε τι προτείνω από τροπολογίες. Στην τροπολογία 4 λέω ότι να συμπεριληφθεί και η εξαγωγή και μεταφορά στις δραστηριότητες των εξορρυκτικών εταιριών. Όχι μόνο η ανακάλυψη κοιτασμάτων και η ίδια η εξόρυξη, αλλά και η μεταφορά και η εξαγωγή του. Γιατί αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις χώρες αυτές. Στην τροπολογία 5 δίνω έναν ορισμό περί του τι εστί σχέδιο παραγωγικό. Για την Κομισιόν το κάθε παραγωγικό σχέδιο πρέπει να αποκαλύπτει όλες του τις λεπτομέρειες γιατί έτσι είναι πιο ακριβείς οι πληροφορίες για τις επιτόπου δραστηριότητες και όχι μόνο για τα γενικά στοιχεία για ολόκληρη τη χώρα. Ανησυχώ όμως μήπως ο ορισμός αυτός της Κομισιόν δεν επιτρέψει στις εταιρείε να εφαρμόζουν διαφορετικούς ορισμούς ανάλογα με τη διαχειριστική των δομή. Και γι' αυτό να υπάρχει περίπτωση να μην είναι λειτουργικός ο ορισμός, να μην είναι συγκρίσιμα τα παρόμοια στοιχεία. Προτείνω λοιπόν να ορίζουμε το κάθε project ως οποιαδήποτε νομική συμφωνία που δίνει δικαίωμα φορολόγησης της εταιρείας στη χώρα όπου λειτουργεί. Όπου υπάρχει διαφορετική βάση, τότε θα αλλάζουν και το τρόπος πληροφόρησης. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η εκμετάλλευση της ξυλίας και οι εξορίξεις καθορίζονται ρητά γεωγραφικά. Οι συμφωνίες δηλαδή αφορούν συγκεκριμένες περιοχές. Α, το καλό με αυτόν τον ορισμό είναι ότι σε τέτοιες χώρες ή σε χώρες όπου δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα θα δίνεται η ευελιξία να επι... γίνονται πληρωμές σε διαφορετική βάση. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω έναν ορισμό που να λειτουργεί και για τις χώρες με πολλούς πόρους αλλά που είναι πτωχές και για χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία που δεν ισχύουν οι προηγούμενες συνθήκες. Άρα ο ορισμός λειτουργεί παντού. Στην τροπολογία 69 καλύπτω ορισμένα θέματα που αφορούν το εύρος των πληρωμών. Προτείνω δηλαδή οι αναφορές που γίνονται χώρα με χώρα να διευρυνθούν για να συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς και όχι μόνο τις εξορρυκτικές βιομηχανίες. Και αυτό το λέω μετά από συζητήσεις με τους σκιώδεις όλων των πολιτικών ομάδων. Γιατί κατάλαβα ότι σε πολλές πολιτικές ομάδες υπάρχει άποψη ότι ή δίνεται εδώ η ευκαιρία διεύρυνσης του ορισμού. Παραμένω λοιπόν στοχευμένη στη σημασία της υλοτομίας και των εξορίξεων, αλλά θα ήθελα να ανταποκριθώ και σε αυτά που μου ζητούν οι συνάδελφοι, τον ευρύτερο αυτό ορισμό δηλαδή. Ελπίζω και εσείς να το εγκρίνετε κυρία Πρόεδρε γιατί θυμάμαι ότι στην έκθεσή σας για το 2011 για τη φορολογία και την ανάπτυξη είπατε ότι οι μελέτες χώρα με χώρα έχουν μεγάλη σημασία για τις ψωρικτικές εταιρείε, αλλά θυμίζατε ότι το ίδιο θα ωφέλιμα θα ήταν αυτό και για τους επενδυτές και επενδύτριες. Μάλιστα για να αποφευθεί η φοροδιαφύγη χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες χώρα με τη χώρα. Γι' αυτό προτείνω επίσης κι άλλες λεπτομέρειες να δοθούν πέραν από αυτές που ορίζει η Κομισιόν. Η αποκάλυψη των πληρωμών δεν αρκεί για να φανεί αν πληρώνουν σωστά τους φόρους τους οι εταιρείε. Ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ανησυχεί τις αναπτυσσόμενες χώρες και ο ΣΑ συμφωνεί ότι η φοροδιαφυγή κοστίζει πολλά, πολύ περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι παίρνουν και ως βοήθεια. Γι' αυτό στην τροπολογία 18 λέω οι αναφορές να συμπεριλαμβάνουν και πρόσθετε οικονομικές πληροφορίες χώρα με χώρα, δηλαδή και τις ποσότητες και τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων κλπ πολλές παραπάνω λεπτομέρειες για να μην αφήσουμε κανένα παραθυράκι. Πιστεύω όμως ότι το ουσιοδέστερο απ' όλα είναι η ανάλυση ανασχέδιο. Και ιδιαίτερα για την υλοτομία και τις εξορίξεις πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αναφορές θα γίνονται με βάση σχέδιο το σχέδιο. Και αυτό το λέω σαφώς στην τροπολογία 9. Οι αναφορές αυτών των πληροφοριών από τις εταιρείες ε, λέω να γίνονται με τακτά ενιάφσια, δηλαδή ετήσια βάση. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους επενδυτές και επενδύτριες. Και κάνα δυο άλλα που θέλω να τονίσω. τονίσω. Στην τροπολογία 17 μιλάω για το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να αποκαλύπτουν τις πληρωμές τους οι εταιρείε. Έχει συζητηθεί πολύ από διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου και προτείνω οι πληρωμές να γνωστοποιούνται εάν κάποια πληρωμή ή ένα σύνολο πληρωμών ιδιού τύπου αν έρχεται σε ποσό άνω των 15.000 ευρώ. Αυτό είναι πολύ χαμηλό όριο σε σύγκριση με αυτά που συζητούν άλλες επιτροπές, αλλά όσοι γνωρίζουμε την κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες θα γνωρίζουν ότι τα 15.000 ευρώ είναι πολλά λεφτά αφού μιλάμε για προγράμματα σε τοπικές κοινότητες, στην Αφρική, και ότι αυτό το ποσό αρκεί για να δημιουργήσει τρομερή διαφθορά αν δεν το, αν δεν αντιμετωπίσουμε... αν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά. Γι' αυτό το βάζω εδώ. Βέβαια θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις άλλες επιτροπές για το ποσόν που μπορεί να έχουν ορισμένε διαφωνίες. Και τέλος, για το θέμα των εξαιρέσεων. Η Κομισιόν προτείνει οι εταιρείε να εξαιρούνται από την αναφορά των στοιχείων σε οποιαδήποτε χώρα της οποίας το ποινικό δίκαιο απαγορεύει τέτοιου είδου αποκαλύψεις. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που δείχνουν ότι δεν δείχνει τίποτα ότι υπάρχουν τέτοιοι νόμοι σε οποιαδήποτε χώρα. Και άρα εδώ πρόκειται για όθηση, για περαιτέρω διαφθορά. Οι χώρες δηλαδή που δεν έχουν τέτοιους νόμους θα τους δημιουργήσουν αμέσως με αυτή την ευκαιρία. Δεν πρέπει να δώσουμε τέτοια όθηση. Και τελικότατα ευχαριστώ τους Κιώδης από τις άλλες ομάδες διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και με βοήθησαν πάρα πολύ οι συναντήσεις μας. Ελπίζω δεν να συνεχίσουμε τέτοιου είδους συνεργασία που με βοήθησε τόσο πολύ επαναλαμβάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ιζαμπέλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Φιώνα Χόλ επίσης για αυτήν τις εξαίρετες ε, εκθέσεις. Η κυρία Σαρτζετίνη είναι σκιώδης ε, από τους Πράσινους, αλλά μιλάει στην Κωνσταντινούπολη σήμερα σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη για την μετανάστευση και εγώ την αντικαθιστώ εδώ εκ μέρους των Πρασίνων. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Χόλ για την εξαίρετη εκθεσή της που υποστηρίζουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Συμφωνούμε για το ότι η αρχή ε, σχέδιο προς σχέδιο αποτελεί στοιχείο κλειδί για αποτελεσματική διαφάνεια και ότι είναι ο μόνος ο τρόπος ώστε οι τοπικές κοινότητες που ζουν κοντά σε τέτοια προγράμματα να αντιλαμβάνονται πόσος πλούτος δημιουργείται από τα προγράμματα αυτά και πού καταλήγει. Η κυρία Χόλ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά προσθέτοντας κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τους ορισμούς των προγραμμάτων αυτών, των σχεδίων αυτών, για να μην υπάρχουν κενά και παραθυράκια. Χαιρόμαστε επίση που η συγκήτρια θέλει να αφαιρέσει την ρήτρα εξαιρέσεων από την πρόταση τη Επιτροπή. Η πράξη τα Φρανκ δεν νομίζουμε ότι βοηθάει όταν έχουμε μια τόσο σημαντική νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει κίνητρα προς μια τέτοια στραβή κατεύθυνση όπως πολύ σωστά τόνισε και η κυρία Χόλ. Στηρίζουμε επίσης και την προσέγγιση της εισηγητρίας που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ε, κάποια, κάποιες οροφές ποσοτικές μέσω των κατεξουδότηση πράξεων. Πιστεύουμε επίσης ότι το όριο πρέπει να είναι χαμηλό, όπως προτείνει και η συγκήτρια. Πρέπει να δούμε την υπόθεση αυτή από την πλευρά των τοπικών κυβερνήσεων, δηλαδή τι θα θεωρούσαν σημαντικό ποσό οι τοπικέ κυβερνήσει. Οι πράσινοι επίσης χαίρονται για αυτά που αναφέρει η κυρία Χόλ όσον αφορά την ε, ε, έκθεση πρωτοβουλίας που έκανε η Πρόεδρός μας, η κυρία Βαζολή, όσον αφορά την φορολόγηση και την ανάπτυξη που έγινε το Μάρτιο, όπου αναφέρεται το θέμα των φορολογικών κερδών, που θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της καταπολέμησης της διαφθοράς. Τώρα το ότι και άλλοι τομείς έχουν ε, εδώ τη σημασία τους. Πράγματι, αυτό το πιστεύω εμείς οι πράσινοι. Εγώ το έχω πει και παλιότερα, για την αλία για παράδειγμα. Γιατί η αλία είναι βέβαια φυσικός πόρος και ένα αγαθό ε, για τον κόσμο από ορισμένε χώρε. Οι κυβερνήσει όμω ε, συχνά αναγκάζονται και δίνουν πρόσβαση στου φυσικού του πόρου σε εκείνου οι οποίοι πληρώνουν καλύτερα. Και το χειρότερο είναι ότι τελικά κανεί δεν ξέρει πόσε φορέ πουλούν την πρόσβα... το δικαίωμα αυτά πρόσβασης στους ίδιους για τους ίδιους πόρους. Δηλαδή λέμε ότι η αλία είναι ανανεώσιμος πόρος, αν όμως υπάρχει υπερβολική εκμετάλλευση, τότε θα έλεγα ότι πρόκειται για εξορρυκτική βιομηχανία και όχι για, μια, για ένα κλάδο που έχει ανανεώσιμου πόρους. Γιατί όταν γίνεται υπερβολική εκμετάλλευση, τότε πάβουν, υπάρχουν και αρκετοί πόροι. Το ίδιο ισχύει και με τα τρόφιμα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι την εισηγήτρια. Μια που προτείνει, αν κατάλαβα καλά, προτείνει ε, να γίνεται αναφορά για κάθε πρόγραμμα χωριστά όσον αφορά την εξοριστική βιομηχανία. Έχουμε τώρα και τις άδειε αλίευσης τώρα που αφορούν ε, στόλους τα ανοιχτά. Κατά τη γνώμη μου, όπως σας είπα, θα ενέπιπτε πάρα πολύ καλά στον ορισμό αυτό της εξοριστικής βιομηχανίας γιατί υπάρχει και το login και στην ε, εξορρυκτική βιομηχανία. Οπότε ρωτάω την εισηγήτρια, πιστεύει ότι θα μπορούσε να ήταν δυνατόν να προσθέσουμε και την αλία στον ορισμό αυτό, εξόριξης. Για να ολοκληρώσω, οι πράσινοι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ε, από την έκθεση αυτή. Συμφωνούν και με την γραμμή της εισηγήτριας. Θα υποβάλουν κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουν κάποια σημεία και για να ε, ζητήσουν και κάποιες διευκρινήσεις. Τέλος, η πρόταση αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές, ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την φοροδιαφυγή. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Στην ε, ε, Αφρική, για παράδειγμα, τα έσοδα από την εξόριξη είναι 6 φορές περισσότερο από ό,τι από την ε, βοήθεια που παίρνουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πείσουμε και του συναδέρφου άλλες επιτροπές και το Κοινοβούλιο ολόκληρο και το Συμβούλιο, ώστε το κείμενο να παραμείνει φιλόδοξο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Θα λάβω και εγώ το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την συγήτρια, την κυρία Φιώνα Χόλ, για το πολύ καλό έργο της. Για το γεγονός ότι διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του κυμπένου σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητε για τα κατόφλια που αναφέρει γιατί αυτό το κατόφλι τώρα συμφωνεί με το κατόφλιο των ε, ενεργειών κατά της λεύκανσης χρημάτων, έχω να σας θέσω ένα ερώτημα. Το κείμενό σας περιλαμβάνει μονάχα τις πληρωμές που γίνονται στις κυβερνήσεις. Μήπως είναι αυτό κάπως περιοριστικό όμως, γιατί υπάρχουν και τοπικές αρχές. Υπάρχουν ε, εταιρείες κρατικές οι οποίες μπορεί να πάρουν πληρωμές Παραδείγματο χάρη στην Καμπόν, στην Ιγυρία υπάρχουν κρατικές εταιρείες οι οποίες έχουν ε, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μπορούν να τύχουν αμέσων πληρωμών. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση, αν θα πρέπει να υπάρχει δήλωση για όλες τις πληρωμές που γίνονται στην κυβέρνηση και στις κρατικές εταιρείες γιατί αλλιώς είναι πολύ εύκολο να παρακάμψει το κείμενο αυτό, γιατί δεν αναφέρει τις πληρωμές που γίνονται σε φυσικά, ε, σε φυσικά πρόσωπα. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντέβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσο ήσασταν απούσα και εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες εδώ πέρα να προχωρήσω τα θέματα της Επιτροπής μας. Είναι πολύ θετικό που σας ξαναβλέπω. Να συγχαρώ την Φιώνα Χόλ για μια θαυμάσια έκθεση. Έχει καταλάβει που βρίσκεται ο πυρήνα των προβλέμων, των προβλημάτων και τα σχόλιά της και οι παρατηρήσεις της είναι ιδιαίτερα ευστοχές. Τώρα κάτι ακόμα. Όταν πηγαίνει κάποια εταιρεία και επενδύσει σε μια αναπτυσσόμενη χώρα κάνουν πολλές φορές αντισταθμιστικές επενδύσεις. Δηλαδή δίνουν μια ε, υπόσχεση στις κυβερνήσεις ότι εκεί που εξορίσουν παραδείγματος χάρη θα δώσουν αντισταθμιστικά ωφέλη με τη μορφή ενός σχολείου, ενός νοσοκομείου κτλ. Έχουν λοιπόν κάποια εξισορρόψη που γίνεται, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε διαφθορά γιατί αντί να χτιστεί ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο, πηγαίνουν τα χρήματα στα θυλάκια κάποιου υπουργού. Θα ήθελα λοιπόν να στήσω από τη Φιώνα να εξετάσει πώς η έννοια των αντισταθμιστικών επενδύσεων μπορεί να ληφθεί υπόψη, ώστε ότι κάνουν μέσα στα πλαίσια αυτά οι πολυεθνικές εταιρείε να καλύπτεται από την ανάγκη της διαφάνειας. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς επιστρέψατε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ως εκπρόσωπο της Σοσιαλιστικής Ομάδας να ευχαριστήσω την κυρία Χολ για τη θαυμασία εκθεσή της. Είναι λοιπόν, <clears throat> ήταν καθήκον του Κοινοβουλίου μας να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα το οποίο το συζητήσαμε διαμακρών στην Επιτροπή μας και είμαι σίγουρο ότι θα ευδοκιμήσει αυτή η έκθεση. Η σοσιαλιστική ομάδα πιστεύει ότι προφανώς θα πρέπει για κάθε σχέδιο να αναφέρουν τις πληρωμές τους οι εταιρείε, αλλά στις τροπολογίες μας υπάρχει και μια βασική ιδέα που νομίζω ότι είναι σημαντική και για αυτή την έκθεση. Είναι ότι θα πρέπει η δημοσίευση αυτών των πληρωμών προς τις δημόσιες αρχές να εξασφαλίσει και μια καλύτερη εικόνα για τη ροή των εσόδων, ώστε η κοινωνία των πολιτών να γνωρίζει τι γίνεται στις χώρες αυτές, τις φτωχέ αυτές χώρες, οι οποίες είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους συνήθως. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μια μεγαλύτερη διαφάνεια να εξασφαλίσουμε και μια καλύτερη ευκυβερνησία στις χώρες αυτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η εκθεσή σας καλύπτει σε μεγάλο βαθμό ένα κενό το οποίο υπήρχε ήδη στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Που εκπροσωπείται από την κυρία Καλίνα Σιμών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Συγήτρια. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς, από την ομάδα που έχει να κάνει με την λογιστική οδηγία, αλλά ασχολούμαστε και με την οδηγία για τη διαφάνεια που εξετάζει τις αναφορές αναχώρα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την έκθεσή σας και για τη δουλειά που έχετε κάνει και για την στήριξη που προσφέρετε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην παραβλέψουμε. Ένα από αυτά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση αυτή προσπαθεί να επικεντρωθεί σε τομεί που δεν είναι ακριβώς ανανεώσιμοι. Γιατί άλλοι που πήραν το λόγο είπαν ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, αλλά επί του παρόντο πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε αυτού του δύο τομεί. Γιατί καλύπτονται και από την νομοθεσία των ΗΠΑ την ε, εξοριστική δηλαδή βιομηχανία, αλλά και την υλοτομία. Τονίζω ότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής αποτελεί προϊόν τεράστιων προσπαθειών ε, που κάναμε για να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην χρηστή διαχείριση και την διαφάνεια, αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε να αποφύγουμε να βάλουμε σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι σε επίπεδο λεπτομεριών αυτές που έχει δώσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν θα έπρεπε να φτάνουν. Ίσως να γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο έχει μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Γι' αυτό θα έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό για να δούμε τι είναι εφικτό σε αυτό το στάδιο. Να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτούς τους δύο τομείς, να αποφύγουμε υπερβολικές προσδοκίες οι οποίες τελικά μπορεί να μην μας οδηγήσουν πουθενά. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αντίσταση αλλά και μεγάλη στήριξη ε, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής. Το θέμα της ε, αποφυγής της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα λογιστικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, πρέπει να ξέρετε. Δεν μπορούμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για φορολογικούς παραδείσους ή άλλες μεθόδους φοροδιαφυγής. Το άλλο που θέλω να πω είναι το θέμα του επίπεδου διακυβέρνησης. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι πληροφορίες να μπορούν να είναι και σε επίπεδα τοπικής επιχείρησης ή ε, τοπικών επιχειρήσεων που παίρνουν τα χρήματα αυτά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινότητες κυρίως. Η προσέγγιση σχέδιο προς σχέδιο είναι μια πολύ καλή. Στο Συμβούλιο ακούστηκαν κάποιες φωνές κατά. Ε, Εμεί θα επιμείνουμε να διατηρηθεί γιατί αποτελεί και τον πυρήνα της πρότασης αυτής. Γιατί έτσι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια και αυτό ακριβώς εμείς επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Η συγκήτρια, κυρία Χολ, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια. Θέλω να επανέλθω σε μερικά σημεία παρακαλώ. Για το θέμα της αλίας. κατανοώ πάρα πολύ καλά γιατί είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο. Για να ξέρουμε τι πληρωμές ε, λαμβάνουν οι διάφορες κυβερνήσεις, ναι. Η πρώτη αντίδρασή μου όμως είναι ότι θα ήταν δύσκολο να το συμπεριλάβουμε στα πλαίσια αυτής εδώ της οδηγίας. Γιατί μιλάμε για πολλές ε, επιχειρήσεις εντός εκτός χρηματιστηρίου και δεν ξέρουμε κατά πόσο η αλία και οι άδειε οι αλλιευτικές πάνε σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Για το θέμα τώρα των πληρωμών στι τοπικές κυβερνήσει, Κάτι πρότισε η κυρία και τον, ο κύριος Ντέβα και ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ, αλλά ε, η κυβέρνηση στον ορισμό του άρθρου 36 λέει η κυβέρνηση σημαίνει κάθε εθνική περιφερειακή τοπική αρχή ενό κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας και περιλαμβάνει και τμήματα, υπηρεσίε ή επιχειρήσει που ελέγχουν οι τοπικοί αυτοί παράγοντες. Πιστεύω ότι υπάρχει κάλυψη εδώ. Διασφαλίζουμε δηλαδή έτσι ότι και οι τοπικές αρχές και οι τοπικές οργανώσεις συμπεριλαμβάνονται εδώ. Ένα άλλο σημείο που θίξατε είναι το θέμα των πληρωμών σε είδος. Και αυτό καλύπτεται από την τροπολογία 9. Είναι ορθό ότι ένα πρόγραμμα που γίνεται ε, μπορεί, εφόσον υπάρξει μια τέτοια ανταλλαγή σε είδος, να οδηγήσει σε διαφθορά. Η τροπολογία 9 το διευκρινίζει και λέει ότι στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων και όλων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην εξορρυκτική βιομηχανία στην υλοτομία, και εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα έργα, προσδιορίζει το ποσό ανατύπω πληρωμής συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών και σε είδος για κάθε τέτοιο έργο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και το συνολικό ποσό πληρωμών ε, κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι έτσι καλύπτονται πάντως είδους πληρωμές, είτε είναι σε είδος είτε όχι. Τέλος. Για την ισορροπία ανάμεσα στην, στην διαφάνεια από τη μια μεριά και ε, την καλή ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων. Πρέπει να ξέρετε ότι έτσι και αλλιώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις το κάνουν ήδη. δίνουν μια έκθεση δηλαδή για τις δαπάνε αυτές. Υπάρχει δηλαδή διαφάνεια. Και όσοι δεν το κάνουν ε, δεν πάνε καλά. αλλά πολλές ακολουθούν σε θελοντική βάση αυτόν τον κανόνα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει πράγματι να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό και ο κανόνας. Ευχαριστώ. Σας ε, μερσώ κυρία Χολ για το έργο αυτό, για τα σχόλιά σας. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι γνωρίζετε ότι η Ιδανική Προεδρία θέλει το νομοθέτημα αυτό να εγκριθεί πριν από το τέλος της, ε, του εξαμήνου της Προεδρίας της και γι' αυτό θα ψηφίσουμε στις 4 Ιουνίου και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι αύριο το μεσημέρι. Και τώρα προχωρούμε. Το επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας τέσσερα σημαντικά, τέσσερις σημαντικές γνωμοδοτήσεις έχουμε για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ένας μηχανισμός που έχει να κάνει με, το, με την γειτονία, το μέσο σταθερότητος, το μέσο συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και αυτό για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τέσσερα αυτά θέματα θα τα αντιμετωπίσουμε αλληλοδιαδόχως. Ξεκινάμε με την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Ντέβα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο σχέδιο γνωμοδότησής μου για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μέσο προτείνω στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πέντε μονάχα και έχουν σαν στόχο οι τροπολογίε αυτέ να βελτιώσουν τη διατύπωση και τη σχέση μεταξύ ανακουφιστική βοήθεια βοήθειας, και ανάπτυξη. Και επίση αναφέρονται στο στόχο τη μείωση της ένδυα. Όλα αυτά συνάδουν με τη νομική βάση που επέλεξε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το ρόλο της δημιουργίας πλούτου που για μένα δεν είναι διαφορετικό από το στόχο μείωση της ένδυα. Δεν μου φαίνεται λογικό να μιλάμε για μείωση της ένδυας χωρίς δημιουργία πλούτου. Πώς αλλιώς μπορεί να εξασφαλίσει κανείς τη μείωση της ένδυας. Μετά από τις άτυπες συνεδριάσεις που έχουν οργανιστεί από τη γραμματεία της ε, ΑΦΕΤ με τη δική μας γραμματεία, νομίζω ότι μια τέτοια μινιμαλιστική αντιμετώπιση που βασίζεται μόνο σε μερικές τροπολογίες, αλλά που αντιμετωπίζει τα κέρια θέματα, ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν να γίνουν δεκτές οι απόψεις μας μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Να σας παρουσιάσω τώρα εν συντομία το, το περιεχόμενο των τροπολογιών μου. Η τροπολογία 1 για το άρθρο 1 του σχεδίου αυτού έχει σαν στόχο να προσθέσει την μείωση της ένδυας μέσα στα πλαίσια της ε, πρότασης της Κομισιόν. Οι τροπολογίες 2, 3 αλλά και 4 για τα άρθρα 2 και 7 έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν τη σύνδεση μεταξύ της μείωσης της ένδυας και της ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας και τη μετάβαση από την έκτακτη ανακουφιστική βοήθεια μετά από μια κρίση ή καταστροφή μέχρι και τη μακροχρόνια αναπτυξιακή βοήθεια. Τονίζουν λοιπόν αυτή τη σύνδεση και τονίζουν και τον ρόλο της δημιουργίας πλούτου για να αντιμετωπιστεί η ένδια. Η τροπολογία 5 στο άρθρο 20. Τεχνική αλλά σημαντική. Η Κομισιόν δεν είχε ημερομηνίε εκπνοής για τα μέσα αυτά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ημερομηνίε που λήγουν αυτά τα εργαλεία. Και εδώ αναφέρεται 31 Δεκεμβρίου 2020. Θα ήθελα φυσικά να ακούσω και τις απόψεις των άλλων συναδέλφων για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Όπως ξέρετε, έχουμε επικρίνει την ε, νοοτροπία more for more, πιο πολλά και για πιο πολλά, και το κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς. Συζητάμε λοιπόν για αυτό το θέμα, αλλά συγχρόνως πρέπει να αντιμετωπίσουμε γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν να ακούσω την άποψή σας για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Νόρμπερ Νόιστερ έχει το λόγο τώρα. τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι και εγώ που σας ξαναβλέπω στην Επιτροπή μας για την γνωμοδότηση του κυρίου Ντέβα. Εξ ονόματος της ομάδας μου, εγώ μπορώ να συνενέσω απόλυτα. Έχουμε βέβαια να αντιμετωπίσουμε πολλές τεχνικές έννοιες που θα πρέπει να τις ε, αντιμετωπίσουμε σωστά, ώστε στο μέλλον να μπορεί η βοήθειά μας να ε, εφαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα στο μέλλον από ό,τι τώρα. Αυτό είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα ιδίως ε, σε ό,τι αφορά την σχέση γειτονία μα με την νότια όχθη τη Μεσογείου και τον αραβικό κόσμο. Εκεί τα άτομα είναι αδίμονα και περιμένουν συγκεκριμένε ενέργειες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να μας δώσουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο λειτουργικοί και προσαρμοσμένοι στι τοπικέ συνθήκε. Το σύνθημα «more for more» Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε βέβαια καταρχήν, ότι άμα είναι καλή εξέλιξη θα έχει ακόμα και ταχύτερη υποστήριξη, αλλά σημαίνει επίσης και less for less, δηλαδή όταν καθυστερεί η ανάπτυξη δεν θα υπάρχει παροχή πόρων. Αυτό όμως πρέπει να το συζητήσουμε γιατί δεν πρέπει να είναι ένα πρόσχημα για να αποσύσουμε την ευθύνη που έχουμε να βοηθήσουμε τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι είναι σημαντικό να συνδέσουμε την στρατηγική γειτονία με την νότια όχθη της Μεσογείου με τις σχέσεις Ευρώπης με την Αφρική και ιδίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και μέσα σε γενικότερες παγκόσμιες πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον. Αυτό είναι μια ευκαιρία και για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουμε και περαιτέρω συμμάχους όταν πρόκειται για την επίτευξη λύσεων για την κλιματική αλλαγή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών μεταξύ της άμεσης βοήθειας, της ανοικοδόμησης και της αναπτυξιακής βοήθειας. Και στον τομέα αυτό θα πρέπει η μεσοπρόθεσμη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί. Αναφέρεται η κοινωνία των πολιτών. Εγώ με την προηγούμενη εβδομάδα στον διαρθρωμένο διάλογο και άκουσα εκεί πολλές ε, επικρίσεις από τις τοπικές αρχές, οι οποίες πολλές φορές πιστεύουν ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνία των πολιτών από ό,τι στις τοπικές αρχές. Ναι, μεν χρειάζεται να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά παράλληλα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις τοπικές αρχές, γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε την καλύτερη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε αποκέντρωση, δημοκρατικοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία της βοήθειας. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό από τη δική μας οπτική γωνία είναι ότι σαν Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια για το εργαλείο της δημοκρατίας να μην αποδοθούν για τους σκοπούς του μέσου γειτονίας και τέλος οι τροπολογίες του κυρίου Ντέβα είναι πραγματικά τόσο ρεαλιστικές που θα υποστηριχθούν και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Από τη δική μας πλευρά θα κατατεθεί μια τροπολογία ακόμα για το άρθρο όταν τονίζουμε για την ανάγκη της αηφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και την προστασία των πόρων ποσίμου ύδατος, όπως επίσης και την προστασία των θάλασσων. Και χαίρομαι και πάλι για την αξία αυτής της έκθεσης. Ο κύριος Γκέρανς. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με μια κοινοτοπία. Ο κύριος Ντέβα έκανε καλή έκθεση. Έχει γίνει πια κοινοτοπία αυτό γιατί δεν μπορεί να κάνει κακή έκθεση, είναι ανίκανος. Ή μάλλον δεν είπα ανίκανος γενικά, ανίκανος να κάνει κακή έκθεση, να μην παρεξηγούμεθα εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα μετά από αυτά που είπε ο κύριος Νόιζερ για το DCI, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε από εκεί λεφτά για να χρηματοδοτήσουμε άλλα προγράμματα. Δεν θέλουμε να αυξομοιώσουμε τα διάφορα προγράμματα για να μην επωφεληθεί ας πούμε ο έρασμος για όλους και όλες. Πάντως από κάπου πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Για λόγους δε σαφήνειας θα ήθελα να μου πείτε τι τμήμα θα δοθεί για, σε αναπτυξιακούς, για αναπτυξιακούς στόχους. Η Κομισιόν μήπως μπορεί να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια ένδειξη ποσοστιαία τι θα χορηγηθεί για αναπτυξιακά ως βοήθεια. Aussi euh, aux propositions que je vais faire dans mon rapport sur le futur agenda de développement. Γιατί πρέπει να το ξέρουμε αυτό και για το μέλλον. Και σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά τον φίλο μας τον Ντέβα. La parole est à la commission. Η commission, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Ανδρέας Ιακώβ. Όχι, Άντριους, Άντριους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άντριου Τζέικομς από την ΔΕΒΚΟ της Κομισιόν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεση του καθώς και το σύνολο των μελών που εξεφράστησαν και σχολίασαν. Πρώτον, για το θέμα της μείωσης καταπολέμησης της ανέχειας. Επιβεβαιώνει, όπως ξέρετε, έχει αναλάβει τη δέσμευση να παίξει καθοδηγητικό ρόλο για την απάλληψη της ανέχειας παγκοσμίω. και γι' αυτόν τον λόγο είπαμε να υπάρξουν και να δοθούν και κονδύλια στοχευμένα σε αυτό ακριβώς το στόχο όπως το DCI, η συνεργασία για την ανάπτυξη και το ίδιο το αναπτυξιακό ταμείο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για όλα αυτά τα εργαλεία και μέσα και προχωρούμε και με το Συμβούλιο και με σας. Ως προς τη γειτονία και την, το νέο αυτό εργαλείο γειτονία. Η μείωση της ανέχειας είναι επίσης πολύ σημαντικός του στόχος μεταξύ άλλων και το αναφέραμε στο άρθρο 2, δέλτα. Αλλά η μείωση της ανέχειας δεν είναι ο μόνος στόχος μας γιατί οι χώρες της γειτονίας έχουν πολλές ιδιαιτερότητες και ειδικέ ανάγκες που πρέπει και αυτές να αντιμετωπιστούν και πέρα από την απάλληψη της ανέχειας. Όπως είπατε, το άρθρο 21 της συνθήκης καθορίζει τους γενικούς στόχους της Ένωσης και των εξωτερικών αυτής σχέσεων και προσδιορίζει την προώθηση βιώσιμης οικονομίας με ανάπτυξη που δεν βλάπτει το περιβάλλον και απαλήφει την ανέχεια. Όσο για το εργαλείο γειτονία, το άρθρο 1 του σχεδίου ΕΝΗ, ENI, αναφέρεται παραπέμπει επίσης στη συνθήκη που μιλάει για δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας. Αυτό είναι η βάση όλης μας της πολιτικής. Για τις τροπολογίες σας προς το 2 νομίζω ότι αυτά που προτείνετε ήδη εννοούνται, υπονοούνται από το κείμενο ως έχει. Κατά την διατύπωση του, τη σύνταξή του και τις συζητήσεις που είχαμε με, προς αυτό με το Συμβούλιο προσπαθήσαμε να μην το παραφορτώσουμε με στόχους. Βέβαια η δημιουργία πλούτου είναι από τους σημαντικότερους αλλά προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των στόχων για να μην αναφέρονται σελίδες επί σελίδων στόχων. Γιατί ένας τέτοιος κατάλογος δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι εξονυχιστικός. Για το 7 θεωρούμε ότι μπορεί όντως να πρέπει εδώ να μιλήσουμε και για τη στήριξη μετά από τις κρίσεις και για την οικοδόμηση της αντίστασης σε κρίσεις των ωφελουμένων και όχι μόνο την αντιμετώπιση των κρίσεων. Τέτοια προγράμματα θέλουμε να προτείνουμε και για τη Λιβύη, αλλά πρέπει να προσέξουμε νομίζουμε στη διατύπωση που αφορά τις μακρόπνοες ε, αναπτυξιακές δραστηριότητες, γιατί πολλές φορές σε ορισμένες χώρες η αντιμετώπιση των κρίσεων δεν είναι αναγκαστικά και σε περισσότερη ανάπτυξη, όπως παραδείγματος χάρη στη Λιβύη, όπου θα υπάρξει μακρόπονο ή μακροπρόθεσμη στήριξη για την ανάπτυξη και όχι μόνο για την αντιμετώπιση. Τέλος, για την ε, προθεσμία που προβλέπεται για την οδηγία, αυτό είναι κάτι οριζόντιο που αφορά όλες, όλα τα σχέδια, κανονισμών μάλλον, όχι οδηγία, Πρέπει να το ξαναδούμε, να δούμε ξαναδούμε αυτή την τροπολογία για να συνδυαστεί και με τα υπόλοιπα εργαλεία και κανονισμούς. Μας ανησυχεί το μήπως αν βάλουμε καταληκτική ημερομηνία την βάλουμε νωρίτερα από την λήξη των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να δούμε όλα τα προγράμματα πώς προχωρούν και ποια θα ήταν μια ρεαλιστική νομική καταληκτική ημερομηνία. Τέλος. Ε, Για την λεγόμενη «dacability» θα επανέλθω επ' αυτού άλλη φορά γιατί ακόμα το εξετάζουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξανά ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν σημαντικά πράγματα. Το more for more και less for less είναι κάτι που είναι πολύ σωστός τρόπος για διάθεση κινήτρων, αλλά το less for less δεν λειτουργεί. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί αλλιώς μπορεί να καταλήξουμε στην απόλυτη φτώχεια ενός πληθυσμού. Μπορεί για ορισμένες χώρες που δεν αναγνωρίζουν τους δικούς μας κανόνες και κανονισμούς για την εύνομη τάξη, τη δημοκρατία κτλ. να δικαιολογείται. Αλλά αν εφαρμόσουμε την αρχή λιγότερα για λιγότερα δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Μπορεί να μην υπάρχει όριο για το παραπάνω για παραπάνω, αλλά για το λιγότερο για λιγότερα υπάρχει. Ο Τσάρλς είναι πολύ γενναιόδωρος προς εμένα, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω εγώ ιδιαίτερα τη γραμματεία μας, που με βοήθησε ιδιαίτερα για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης και πρέπει να το αναγνωρίσω. Νομίζω ότι είναι γελίο, αν μου το επιτρέπετε, η Κομισιό να μας λέει ότι δεν υπάρχει τρόπος, χώρος να μειωθεί ανέχεια και να αυξηθεί ο πλούτος. Αν δούμε τα πράγματα σφαιρικά, έχουμε περίπου 60 δισεκατομμύρια το χρόνο για το στόχο αυτόν. Και αυτά τα 60 δισεκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε σε ένα δισεκατομμύριο περίπου ανθρώπους. Δεν χρειάζεται κανένας φοβερός μαθηματικός για να καταλάβει ότι για ένα δισεκατομμύριο αν διαθέτουμε 60 δισεκατομμύρια, τότε τους δίνουμε 60 ευρώ τον καθένα το χρόνο. Δηλαδή 16 λεπτά την ημέρα. Μπορεί κανείς εδώ να μας πει ότι με τέτοια ποσά θα απαλείψουμε την ανέχεια με 16 λεπτά την ημέρα που θα διαθέτουμε στους φτωχούς. Όχι βέβαια. βέβαια. Ας μιλήσουμε λοιπόν μάλλον για τη δημιουργία πλούτου. Αυτά τα 16 λεπτά δεν κάνουν τίποτα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν οι δομές που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους αυτούς να κερδίσουν 1,6 με 2 ευρώ την ημέρα. Όχι απλώς να τους δωρήσουμε 16 λεπτά, γιατί αυτό δεν θα μειώσει καθόλου την ανέχεια. Να μην εξισώνουμε λοιπόν τις δωρεές με μείωση της ανέχειας. Δεν έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Το μόνος τρόπος είναι η δημιουργία πλούτου. Όχι 16 λεπτών, αλλά το τριπλάσιο και το τετραπλάσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η Τετάρτη, 30 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση αυτή αυτή στις 19 Ιουνίου στη συνεδρίασή μας και η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει την δικιά της έκθεση στις 9 Ιουλίου. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Δημιουργία ενός μέσου εταιρικής σχέσης για συνεργασία με τρίτες χώρες. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Κυρία Σαλώμα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησής σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην Επιτροπή μας, κυρία Πρόεδρε, μετά από ένα στάδιο τόσο ταραγμένο στην πολιτική σας ζωή. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι ενώ εσείς αγωνιζόσασταν για τις ιδέες σας στην προεκλογική εκστρατεία της Γαλλίας σας, ε, αντικατέστησε η κυρία Στρίφλερ, η οποία έδειξε μια μεγάλη θεσμική πίστη απέναντι στην Επιτροπή αυτή. Οπότε συγχαρητήρια και στις δυο σας. Η γνωμοδότηση που ετοίμασα και που παρουσιάζω ξεκινάει από ένα αρχικό σημείο. Αναγνωρίζει το ότι, όπως ξέρετε, υπήρχε ένα άλλο μέσο που αντικαταστάθηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι στην ονομασία υπάρχει μια αλλαγή και στο είδος του μέσου. Το 2000, μέχρι το 2013 είχαμε αυτό που ονομάζαμε μέσο για τη συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες και λοιπές χώρες υψηλού εισοδήματος. Τώρα Προσπαθούμε με τη γνωμοδότηση αυτή να αλλάξουμε τα πράγματα και θα ονομάζεται Μέσο εταιρικής σχέσης. Υπάρχουν ε, διάφορες σχέσεις πολιτικές, εμπορικές, ε, οικονομικές που έχουμε και μας βοηθάει το μέσο αυτό. Από το 2007 που άρχισε το προηγούμενο μέσο και 2014 που θα ξεκινήσει το νέο, έχουν συμβεί πολλά πράγματα στον κόσμο. Το πιο σημαντικό, δίχως άλλο, είναι ότι αναδύονται νέες οικονομίες, με ιδιαίτερη ισχύ όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, αλλά και άλλες, που καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις αλλά και στις πολιτικές σχέσεις και στρατηγική σημασία σχέσεις στον κόσμο. Πρόκειται δηλαδή για παράγοντες σημαντικούς γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει κάθε συμφέρον να ε, συνδεθεί μαζί τους και όχι μόνο στο εμπορικό επίπεδο, ούτε μόνο στο επίπεδο της ανάπτυξης. Όλα αυτά τα χρόνια επίσης η οικονομική κρίση είχε το δικό της αντίκτυπο η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και επηρεάζεται βέβαια και η αναπτυξιακή μας πολιτική από αυτό. Την ίδια εποχή άλλαξαν και αλλάζουν κάποιες από τις γενικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ανά το κόσμο. Μειώθηκε κάπω η ανησυχία για τις κλιματικέ αλλαγέ, λαμβάνοντα υπόψη. Και όταν λέω ότι μειώθηκε, θα έλεγα μειώθηκε η ένταση με την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικέ αλλαγέ, γιατί κάποιες χώρες έχουν βρει ως άλοθη την οικονομική κρίση για να επιβραδύνουν τις προσπάθειε που κάνουν σε αυτό το τομέα. Άλλαξε επίση κάπω και η κατεύθυνση των μεταναστευτικών ροών. Και αυξήθηκε κατά πολύ η ανησυχία όσον αφορά την επισητιστική ασφάλεια και την διατροφή στον κόσμο. Από αυτή την οπτική γωνία λοιπόν, αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο εμπόριο. Εξωτερικές σχέσεις επίσης. Γιατί, γιατί θέλει μέσα από αυτό το μέσο εταιρική σχέση να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 μέσω διμερών συνεργασιών, περιφερειακών συνεργασιών ή και διαπεριφερειακών. Θέλει να βελτιώσει επίσης την πρόσβαση στις αγορές, να αναπτύξει νέες δυνατότητες επενδυτικές και επιχειρηματικές, κάτι το οποίο φαντάζομαι ικανοποιεί ιδιαίτερα και τον κύριο Ντέβα η ανάπτυξη αυτή εμπορικών ευκαιριών και επιχειρηματικών. Το όλο που κάνει είναι ότι προωθεί την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο, από κάθε άποψη. Η στάση αυτή και η θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι λογική, είναι και η θέση που θα υποστηρίξουμε και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, αλλά και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εμείς λοιπόν, τι μένει να κάνουμε, πρέπει να προσθέσουμε την αναπτυξιακή διάσταση σε αυτήν την καινοτομία που γίνεται για τον μέσο. Και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ βασικό να εισακάγουμε κάποια στοιχεία από την οπτική γωνία ακριβώ της ανάπτυξης προκειμένου να συμπληρώσουμε την ε, θέση αυτή για οικονομική και εμπορική συνεργασία. Πώς, με τι. Πρώτα απ' όλα, η γνωμοδότηση λαμβάνει υπόψη ότι οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους και μάλιστα ορισμένες έχουν, που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό οικονομικά. Η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία για παράδειγμα έχουν βγάλει από τη φτώχεια πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Εκατοντάδες θα έλεγα εκατομμύρια ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά στις χώρες αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια φτωχοί. Και η κατανομή βέβαια δεν είναι καθόλου ισόρροπη εξαρτάται από το φύλλο, από την γενιά, από την γεωγραφική τοποθεσία όπου βρίσκονται, από τη μόρφωση και πολλά άλλα. Συνεπώς, τη στιγμή που θέλουμε να εισαγάγουμε την προοπτική, την αναπτυξιακή στις δικές μας εμπορικές σχέσεις, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε αυτές τις χώρες το μέσο εισόδημα μπορεί να έχει αυξηθεί πολύ, κατά μεσό όρο δηλαδή, παρόλα αυτά υπάρχουν θύλακες τρομερής φτώχειας. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε δηλαδή τι ανισότητε. Δεύτερον, συνοχή. Πιστεύουμε ότι ακριβώς επειδή μιλάμε κυρίω για εμπορικέ σχέσεις, είναι πολύ βασικό να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση με αρχές ε, δικέ μα κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει και συνοχή με άλλους μηχανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Μια άλλη πτυχή που συμπεριλαμβάνεται στη γνωμοδότησή μου είναι η ανάγκη να ελέγξουμε, να παρακολουθήσουμε την λειτουργία των μέτρων που υιοθετούνται. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται και συγχρόνως θα εκφράζει την άποψή του για την πρακτική που ακολουθούμε. Το επόμενο, δεδομένου ότι υπάρχει κάτι που υποστηρίζουμε πάρα πολύ, δηλαδή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να φροντίσουμε η συμμετοχή αυτή του ιδιωτικού τομέα να συνάδει με την πρόθεση των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλων βασικών αρχών που στηρίζει παραδοσιακά η Επιτροπή μας. Τέλος, υπογραμμίζω ότι σε διάφορους τομείς πρέπει να στηρίξουμε την προστιθέμενη αξία που είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον από τις δράσεις των χωρών μελών. Δηλαδή είναι προτιμότερο μια δράση να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά να γίνεται επιμέρους στις διάφορες χώρες μέλη. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία. Συνεπώς προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή μάλλον Εξωτερικών Υποθέσεων να συμφωνήσει με την αρχή αυτή της πρόσθετης αξίας. Γιατί είναι μια πρόσθετη αξία η οποία αποδεικνύεται κάθε φορά όταν αξιολογούμε τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ένα σημείο στη γνωμοδότησή μου είναι ότι πρέπει να μάθουμε, να πάρουμε μαθήματα από το ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ώστε να φροντίσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί κάθε φορά που θα χρησιμοποιούμε αυτό το νέο μέσο. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Το μέσο αυτό λαμβάνει έναν κάπως διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με αυτό που αντικαθιστά. Επικεντρώνεται κυρίως στο εμπόριο, κυρίως στις εξωτερικές σχέσεις και νομίζω ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να ζητήσει να προσθεθούν κάποια στοιχεία που ενδιαφέρουν τη δικιά μας την Επιτροπή Εξού και προτείνουμε κάποιες τροπολογίες σε διάφορα άρθρα του μέσου. Ευχαριστώ. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ επειδή έχω πίεση χρόνου επειδή στις 6.30 πρέπει να είμαι στο Λουξεμβούργο για μια στόκυλη τράπεζα, δεν θα μπορέσω να περιμένω την απάντηση που θα μου δώσει η Κομισιόν. Μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Γκερέρο. Να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ, ότι χρειάζεται μια συνεχής εξέταση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από αυτό το μέσο. Βεβαίω. Εγώ όμως θα θέλω να ξέρω, δεδομένου του του ότι η συζήτηση που κάνουμε τώρα συνδέεται άμεσα με τη διαφοροποίηση που προτείνει η Κομισιόν στα πλαίσια της μελλοντική ατζέντα, ποιο θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα όταν πρέπει να γίνει μια εκταμίευση από το νέο μέσο εταιρικής σχέσης. Αν έχω καταλάβει σωστά, και ήδη εγώ θέλω να τα εντάξω αυτά στη μελλοντική μου έκθεση για τον φορέα ανάπτυξης, αν έχω καταλάβει καλά η Κομισιόν θα θέσει πέρας στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία με ορισμένες χώρες που έχουν πλέον ενδιάμεσο κατακεφαλής, κατακεφαλής όριμα. Το, για τις εκταμίευσεις τώρα που θα προκύψουν, αυτές οι εκταμίευσεις θα γίνονται στη, υπέρ της πολιτικής ανάπτυξης, μα αυτό θα είναι ενάντιο της αρχής διαφοροποίησης, Δεύτερον, εμείς έχουμε ήδη κάνει μια επισκόπηση, ιδίω στη Λατινική Αμερική, για τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν υποστηριχθεί από το πρόγραμμα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της τωρινής περίοδου χρηματοδότησης, δίνοντας έμφαση στο ότι οι χώρες αυτές δεν θα έπρεπε στο μέλλον ως αναδυόμενες χώρες να υποστηριχθούν από αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν όμως να συμμετέχουν σε μια τριγωνική συνεργασία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο χορηγός και μία αναδυόμενη χώρα θα μπορούσε να είναι πάροχος υπηρεσιών και μια αναδιόμενη ως δικαιούχος των επιδοτήσεων. Μα πώς η Κομισιόν στο μέλλον θέλει να ειναι παροχος υπηρεσιων και μια αλλη αναδιόμενη χωρα ως δικαιουχος των επιδοτησεων μα πως η κομισιον στο μελλον θελει να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα DCI. Ακόμα και αν το χρήμα θα περνά από μια χώρα ενδιαμέσου εισοδήματος, που δεν θα μπορεί να έχει αναπτυξιακή βοήθεια λοιπόν, ποιος θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο μέσα σε μια τέτοια τριγωνική ενέργεια. Αυτό είναι το δεύτερο μου ερώτημα. Και κατά πόσον στο μέλλον και το είχα θέσει εδώ τώρα ερώτημα στην Κομισιόν που δεν μου απάντησε. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο στο μέλλον η Κομισιόν μπορεί να αναλάβει τη δέσμευση να περιορίσει τις χορηγίες προς τις χώρες ενδιάμεσου εισοδήματος σε χορηγίες που αφορούν την τεχνική αρρωγή και μόνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντίβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ενρίκο και τη γνωμοδότησή του και τις απόψεις που διατυπώνει και άκουσα μεγάλη προσοχή όλα αυτά που λέτε. Ο Ενρίκο είπε κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά μέσα σε αυτή την έκθεση για την εταιρική σχέση με αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει μια γενικότερη φιλοσοφία που δεν νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή, η, η ίδια Εκτελεστική Επιτροπή έχει το χρόνο να εξετάσει. Μεταξύ 1960 και 1990 ο αναπτυσσόμενος χώρος δεν έγινε πιο πλούσιος αλλά φτωχότερος. Ο αναπτυσσόμενος χώρος έγινε πιο πλούσιος. Μεταξύ 1990 και 2012 ο αναπτυσσόμενος ε, κόσμος αναπτύχθηκε και έγινε πράγματι πιο πλούσιος και ο αναπτυγμένος κόσμος έγινε φτωχότερος. Κανείς δεν έχει αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους μέσα στα τελευταία 20 χρόνια ανεστράφει η σχετική κάμψη των ε, αναπτυσσομένων χωρών. Αν ή πώς χρησιμοποίησαν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα για να γίνουν πιο πλούσιες. Την προηγούμενη εβδομάδα η Βραζιλία έγινε πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ξεπερνώντα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μα σόκαρε. Τα καταφέραν όμω. Πολλέ χώρε τη Λατινική Αμερική γίνονται τώρα χώρε μεσαίου εισοδήματο. Οι τίγρε τη Ασία έχουν επιτύχει κάτι τέτοιο ήδη στο παρελθόν. Η τελευταία έκθεση του Economist λέει ότι στην Αφρική η οικονομική ανάπτυξη είναι τεράστια και κάποιες αφρικανικές χώρες θα γίνουν αναπτυγμένες και ευμαρείς χώρες. Χώρες μεσαίου εισοδήματος και επέκεινα. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει τις χώρες αυτές να λειτουργούν και τι παθαίνουμε εμείς που δεν έχουμε πια αυτή την οικονομική ανάπτυξη που έχουν οι χώρες οι αναπτυσσόμενες. Αν αλληλεί κανείς αυτή την κατάσταση, κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες συνθήκες, τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν τώρα επιτύχει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Τι διδάγματα αποκομίζουμε από όλα αυτά για να εφαρμόσουμε στις δικές μας χώρες όπου δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι βέβαια μια ευρύτερη συζήτηση από το αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Αλλά είναι μια πρόταση η οποία είναι πράγματι εύστοχη και επίκαιρη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι συντελεστές που οδήγησαν τη Βραζιλία από το να είναι μια πολύ φτωχή χώρα με πάρα πολλέ τένε και δούπολη που έχει ακόμα βέβαια και τώρα να γίνει πλουσιότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι έχει κάνει την Κίνα να βγάλει 300 εκατομμύρια από τη φτώχεια. Τι σπρώχνει την Τανζανία και άλλες χώρες στην Αφρική στο να γίνονται πλούσιες. Σε κάποια μέρα η Τανζανία θα είναι πιο πλούσια από τη Βρετανία, τη Μεγάλη Βρετανία. Τι μηχανισμοί λοιπόν λειτουργούν εκεί, τι παράγοντες είναι αυτοί που έχουν οδηγήσει σε αυτή την εξέλιξη. Τι καταφέραν να πετύχουν σωστό είτε με σχεδιασμό είτε στην τύχη. Δεν ξέρω. Και επομένως με ποιους παράγοντες, με ποιους συντελεστές τα έχουμε κάνει σαλάτα και η Ισπανία έχει το μεγαλύτερο ε, ποσοστό ανεργίας και οικονομική κάμψη και γιατί έχουμε και μηδενική μεγέθυνση στην, ε, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε μια τραπεζική κρίση, αλλά αυτό κανονικά δεν πρέπει να έχει καμιά επίπτωση στην ανάπτυξη. Δεν έχω λοιπόν τις απαντήσεις σε όλα αυτά, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση και άλλες εκθέσεις για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς επηρεάζονται όλα αυτά τα πράγματα και πώς κάπου λειτουργούν τα πράγματα ή όχι. Να το κάνουμε με ένα επιστημονικό τρόπο και θα χαιρόμουν πολύ αν κάποιος στην Επιτροπή μας ή κάποιος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν μπορούσε να κάνει κάποια μελέτη και να εξηγήσει πώς οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα η Βραζιλία από χώρες ζήτουλες στη δεκαετία του 70 και του 80 καταφέραν να είναι πλούσιες χώρες. Τι έγινε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Όσε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να σχολιάσει το μέσο εταιρικής σχέσης. Ο κύριος ΟΕΣΕΣ. Λέγομαι Ελισμάτης από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εργαζόμαστε μαζί με το Μέσο για Εξωτερική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να κάνω, ε, να κάνω μερικά σχόλια για αυτά που είπε ο Πρόεδρος και τα μέλη Τη επιτροπή σας και να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματά σας, χωρί τώρα βέβαια να μπω σε λεπτομέρεια στις τροπολογίες σας, οι οποίες αντανακλούν τις προτεραιότητε τη Επιτροπής σας. Να σα υπενθυμίσω μονάχα τα κύρια σημεία της πρότασης για το εργαλείο εταιρική σχέση που έχει πρότεινει η Κομισιόν για να απαντήσω σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Είναι τμήμα αυτό το μέσο ε, ενό ένα τμήμα ενός πακέτου προτάσεων που εγκρίθηκε από την Επιτροπή και εφαρμόζεται στο γενικότερο πλαίσιο της πολιετούς στρατηγικής στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Το κύριο, η κύρια ψηφίδα αυτού του πλαισίου είναι η εταιρική σχέση στις εξωτερικές σχέσεις που έχει σαν στόχο να προωθήσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Αντίθετα με τα εργαλεία για τις βιομηχανικές χώρες ή το ICIC, αυτό το εργαλείο θα έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και τονίστηκε και από τον εισηγητή ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ευρύτερες στρατηγικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πρόθεση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 κτλ. Γενικά να δώσει υψηλότερο προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το εργαλείο προφανώς θα είναι συμπληρωματικό με το DCI, το εργαλείο για τις αναπτυσσόμενες χώρες μαζί με τους στόχους καταπολέμησης της ένδυας. Θα αντιμετωπίζει όμως θέματα που είναι πέραν της ίδιας της ανάπτυξης με χώρες οι οποίες όπως είπε ο εισηγητής διαδραματίζουν ένα ισχυρό ρόλο στον παγκόσμιο χώρο Επομένως, μαζί με τον DCI, το μέσο αυτό θα προωθήσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να γίνει μέχρι τώρα με την εργαλειομηχανή, με την εργαλειοθήκη μάλλον, που έχει στη διάθεσή τη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να υποστηρίξουμε χώρε που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε πολιτικό διάλογο ο οποίο προωθεί τα κοινά μα συμφέροντα και θεωρούμε ότι το εργαλείο αυτό εταιρική σχέση θα παίξει ένα κομβικό ρόλο υποστήριξη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στρατηγικούς εταίρους της σε εισαγωγικά όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, αλλά και με χώρες όπου είναι δρεωμένη σχέσεις μας όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένε Πολιτείες, Κορέα, η Ιαπωνία κτλ. Το μέσο λοιπόν εταιρική σχέσης δεν είναι υποκατάστατο για την αναπτυξιακή βοήθεια, δεν ακολουθεί τη λογική της ε, βοήθεια τη αρρωγή προ κάποιε χώρε δεν θα μπορούσε παραδείγματο να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει έργα υποδομή και αυτό φαίνεται και από το επίπεδο της χρηματοδότησης που αναφέρεται, που είναι κάτι που είναι ένα τμήμα μονάχα του, αυτών που μπορούν να χρηματοδοτήσουν το DCI, προενταξιακές βοήθειες ή οποιοδήποτε άλλο ευρύτερο εργαλείο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ προσεκτικά το θέμα της προσθέμενης αξίας όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή και από αυτόν που τον ακολούθησε. Είναι σημαντικό όμως να υπερθυμίσουμε σχετικά ότι για τις χώρες μέσου εισοδήματος που ξεπερνάνε πια το επίπεδο της κλασικής αναπτυξιακής βοήθειας, το DCI, και ξέρω ότι θα κοιτάξετε και θα παρεξετάσετε και τον κανονισμό για αυτό το εργαλείο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα και προγράμματα για τα δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν οι χώρες αυτές να είναι επιλέξιμες για αυτά τα προγράμματα. Και επομένως αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η γενική μας αντιμετώπιση και ελπίζω ότι έχω απαντήσει κάποια από τα ερωτήματά σας και προσβλέπουμε στις, ε, στη συμβολή που θα έχετε για, τη γνωμοδότηση, για την ε, έκθεση μάλλον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Γκερέρο, για να ολοκληρώσετε, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Γκερέρο. Ναι, έχω δύο ειδών ερωτήσεις που άκουσα. Πρώτα απ' όλα το θέμα, ε, μια κατηγορία ερωτήσεων απευθύνθηκε βέβαια στην Επιτροπή για το πώς θα προχωρήσει. Και μια άλλη έχει να κάνει με το πώς γίνεται οι χώρες οι λιγότερο αναπτυγμένες αναπτύχθηκαν τόσο πολύ και οι αναπτυγμένες χώρες φτώχυναν σχετικά φτώχυναν. Θα έπρεπε να κάνει κάποιος μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, να δει ε, αυτοί που μένουν πίσω έχουν ε, πολλές φορές φυσικούς πόρους, ε, μεγάλο πληθυσμό και δυνατότητες διεύνησης της αγοράς, οπότε αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τους άλλους οι οποίοι είναι ήδη αναπτυγμένοι. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες του Νότου διαπιστώνουμε ότι τη δεκαετία του 80-90 αναπτύχθηκαν πολλοί, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αναπτύσσονται τώρα, αυτή την εποχή. Είναι δηλαδή ένας προβληματισμός αυτός που έχει βέβαια πολύ νόημα. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο κύριος Ντέβα είναι τι κρίμα που δεν ε, μπορούμε να καθίσουμε και να μελετήσουμε τη διαφοροποιημένη ανάπτυξη στις διάφορες χώρες. Αντιλαμβάνομαι ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ε, Βραζιλία, το να ξεπεράσει η Βραζιλία το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να σημαίνει ένα ανησυχητικό μήνυμα που στέλνεται. Οι ε, Βραζιλιάνοι όμως σε, κατά μέσο όρο ζουν χειρότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε προς το παρόν... Εντάξει, αυτά είχα να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση αυτή στις 15 Μαΐου. Η προθεσμία για κατάθεση για υποβολή πρωτοβουλειών μάλλον είναι στις 15 Μαΐου διορθώνει η Πρόεδρος και θα ψηφίσουμε στις 9, η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει στις 9 Ιουλίου. Εμείς θα ψηφίσουμε στις 4 Ιουνίου. 15 Μαΐου προθεσμία, 4 Ιουνίου ψηφίζουμε εδώ και 9 η ΑΦΕΤ. Τώρα, Κριστιαν, ε, Τελπρέντα είναι εισηγητή για την δημιουργία ενό μέσου σταθερότητο, όμω ε, έχει μείνει στο Βουκουρέστι, είχε ρελμένε υποχρεώσει εκεί. Ο κύριο κύριος Πόγκα όμω θα τον αντικαταστήσει και θα παρουσιάσει αυτό την έκθεση του κυρίου Νταν Πρέντε. Να είσαστε σύντομο, παρακαλώ όμω, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ευχαριστώ κυρία μου. Θα είμαι σύντομο. Θα διαβάσω απλώ τη γνωμοδότηση του συναδέλφου που αντικαθιστώ. Ε, Η δημιουργία ενό εργαλείου σταθερότητα λοιπόν. Το εργαλείο σταθερότητα είναι εργαλείο κλειδί για τη διασφάλιση τη συνεργασία και την ανάπτυξη σε περιπτώσει κρίση. Είναι το εργαλείο τελευταία καταφυγή διότι αυτό χρησιμοποιούμε όταν ξεσπάσει μια τέτοια κρίση που να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα για την ανάπτυξη. Με αυτό το εργαλείο η Ένωση δίνει μια πρώτη βοήθεια σε κατεπίγουσες περιπτώσεις και θέτει τις βάσεις για σχέδια αναπτυξιακά σε τρίτες χώρες. Ο κύριος Πρέντα χαίρεται ιδιαίτερα διότι στην πρόταση αναθεώρησής του η Κομισιόν θέλει να διατηρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του και να αυξηθεί η ευελιξία του που είναι το ιδιαίτερό του χαρακτηριστικό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελε να γίνουν και τρία σχόλια. Ένα, την μελλοντική αύξηση του προπολογισμού του. Δύο, μια επαρκή χρηματοδότηση για μακροπρόθεσμα σχέδια και τρίτον για την επανεισαγωγή του, στο κείμενο των ρητρών που αφορούν μέτρα χρηματοδοτικής εφαρμογής και ένα μηχανισμό αξιολόγησης. Ο κύριος Πρέντα χαιρετίζει την αύξηση του προπολογισμού του EDS κατά πάνω από 40%, πράγμα το οποίο το φέρνει σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ύψους. Αυτό όμως δεν αρκεί παρόλα αυτά για να χρηματοδοτηθούν όλα τα προγράμματα που θα έπρεπε και θα μπορούσε να εφαρμόσει η Ένωση για να συνοδεύει καλύτερα τις πρωτοβουλίες ε, κατάπαυσης σειράξεων σε μεταβατική φάση η Ένωση θα έπρεπε να αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό του εργαλείου αυτού στο μέλλον. Δύο. Με, για την κατανομή τη χρηματοδότηση μεταξύ των διαφόρων συνθετικών του στοιχείων σημειώνει ο κύριος Πρέντα ότι η Κομισιόν προτείνει πάνω από 65% της χρηματοδότησής του να αφιερωθούν σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα για να χρηματοδοτηθούν έτσι καταλήλως οι κατεπίγουσες δράσεις. Αλλά όσο έχει τώρα το κείμενο δεν υπάρχουν ποσοστά ελάχιστα ποσοστά για τις μακροπρόθεσμες δράσεις που είναι και αυτές απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κρίσεων γιατί σε πολλές περιπτώσεις η χρηματοδότηση τέτοιων σχεδίων δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αλέως. Πρόκειται για τα μακροπρόθεσμα λοιπόν σχέδια που θέτουν τις βάσεις για τη συνεργασία και για την ανάπτυξη μετά τις κρίσεις στις τρίτες χώρες. Γι' αυτό ο κ. Πρέντα προτείνει ένα ελάχιστο ποσοστό 20% για τη χρηματοδότηση του EDS, ε, του EDS να αφιερωθεί στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και αυτό το λέει στα άρθρα 4 και 5 και θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από μέτρα που να επιτρέπουν περισσότερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών χρηματοδοτικών εργαλείων για να υπάρξει μια πιο επιτελεσματική χρηματοδότηση και συνέχιση των προγραμμάτων που έχουν ήδη αρχίσει σε προηγούμενη φάση του ίδιας. Εάν οι ρήτρες αυτές δεν μπορέσουν να εγκριθούν εδώ, τότε θεωρεί ο κύριος Πρέντα ότι πρέπει η Επιτροπή μας να, το να ζητήσει κάτι ανάλογο και για την αναθεώρηση άλλων εργαλείων. Και για πιο τεχνικό επίπεδο θεωρεί ότι πρέπει να συμπληρωμάνει το κείμενο και ειδικέ ρήτρε για τα ετήσια προγράμματα δράση και για τα ειδικά μέτρα εφαρμογή. Αν ο σκοπό τη αναθεώρηση είναι να απλοποιηθεί η εφαρμογή του EDS, αυτό δεν πρέπει να γίνει παρόλα αυτά με λιγότερη σαφήνεια και συνέπεια. Θα έπρεπε λοιπόν να επανεισαχθούν εδώ στην πρόταση ειδικέ ρήτρε για την αποτίμηση αξιολόγηση των εγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του EDS και δείκτε να διαμορφωθούν για την εφαρμογή έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του και περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο σα κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ανάγνωσή σας και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για τις παρατηρήσεις της. Ο κύριος Μιχαήλ Ντόιλ. Έτσι μου είπανε. Κανείς δεν είναι Ναι, όχι εγώ είμαι ο Μιχαήλ Ντόιλ. Ένα από, τα, από αυτά που υπόθηκαν ήταν το 20% για τα άρθρα 4 και 5. Εδώ μια αποσαφήνιση. Βλέπω στο κείμενο ότι αναφέρεται στο 20% τουλάχιστον 20% για το άρθρο 4 στην τροπολογία 16. Μπορείτε να μου το εξηγείτε αυτό, ε, αυτή τη διαφορά. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω κανένα συγκεκριμένο θέμα να θίξω. Μόνο αυτό, αν το κατάλαβα καλά. Ευχαριστούμε. Κύριε πόμγα μπορείτε να προσθέσετε τίποτα σε αυτά. Όχι κύριε Πρόεδρε, όχι Καλά. Σα πληροφορώ λοιπόν ότι η διορία κατάθεση τροπολογιών για την κρομοδότηση αυτή λήγει την Τετάρτη 6 Ιουνίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μας στις 19 Ιουνίου και η ΕΠΕΞ θα ψηφίσει στις 10 Ιουλίου. Τώρα το χρηματοδοτικό μηχανισμό για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Ο κύριος Κατσμάρεκ όμως αποσιάζει. Θα περιμένουμε λοιπόν, θα έρθει σίγουρα σε λίγο και περνάμε στη γνωμοδότηση τη δική μου. Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη 67η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΠΕΞ είναι η αρμόδια επί της ουσίας. Παραδοσιακά όμως η ΕΠΕΞ, για την γνωμοδότηση μάλλον, μας δίνει τη δυνατότητα και μας να εκφραστούμε για αναπτυξιακά θέματα. Δίνουμε λοιπόν το λόγο, δίνω το λόγο στον εαυτό μου για να παρουσιάσω αυτή τη γνωμοδότηση. Πρόκειται για τους στόχους της χιλιετίας. Όπως ξέρετε, η τελευταία ημερομηνία είναι το 2015 και οι στόχοι αυτοί τόνισαν ευτυχώς ιδιαίτερα το θέμα της μείωσης της ανέχειας, τη μείωση της θνησιμότητας, της παιδικής θνησιμότητας, την πρόσβαση σε πόσιμο είδωρ κλπ αλλά το 2015 πλησιάζει με ταχαίως και το πρόβλημα τίθεται τι θα κάνουμε για, να, μετά, για μετά το 2015, τι πολιτική όθηση πρέπει να δώσουμε τώρα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι της μίεσης, της ανέχειας ιδιαίτερα. Να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική ορμή που έδωσε που θα δώσει αυτή η 67η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης για να τοποθετηθούμε. Τρεις θέσεις μπορούμε να πάρουμε. Είτε να αναβάλουμε την τελική ημερομηνία, να πούμε ότι ισχύουν μεν οι στόχοι αλλά δεν τους έχουμε πετύχει, δεν θα τους πετύχουμε το 15 και να τους παρατείνουμε. Είτε να κάνουμε κάτι καινούριο με βάση τα επιτευχθέντα, είτε να αλλάξουμε τους στόχους. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να μας πληροφορήσει και είμαι σίγουροι ότι θα το πράξει για την κατάσταση, για την αξιολόγηση που θα κάνει ως προς το τι έχει ήδη επιτευχθεί και ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για την περίοδο μετά το 2015. Υπάρχουν σαφείς ελλείψεις, πρέπει μετά το 2015 να αλλάξουμε λίγο τη μέθοδο εργασίας μας και να έχουμε περισσότερη σύνδεση με την κοινωνία των πολιτών, τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις ίδιες και να δημιουργήσουμε και ένα πάνελ προσωπικότητων σε επίπεδο ΟΗΕ που να αντικατοπτρίζει μια περιφερειακή εξισορρόπηση, εξισορρόπηση μεταξύ των φύλων και να μην αποτελείται μόνον από δωρητάς αλλά και από εκπροσώπους των αναπτυσσομένων χωρών, την, την ερευνητική κοινότητα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσους συντάσσουν τα προγράμματα. Δηλαδή να διευρυνθεί ο, η σύνθεση του. Πρέπει να δώσουμε το λόγο σε όσους δεν τον έχουν ή δεν τον είχαν μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε το ότι εδώ και 50 χρόνια εφαρμόζουμε αναπτυξιακά προγράμματα στη Ζάμπια παραδείγματος χάρη και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το σημαντικό στην κρίση που ζούμε είναι ότι τα κράτη-μέλη μειώνουν συνεχώς τη, τη συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή βοήθεια και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξει τέτοια χρηματοδότηση δεν θα πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Έχουμε αναλάβει την επίσημη δέσμευση να δημιουργήσουμε νέες χρηματοδοτήσεις για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών και οι νέες αυτές χρηματοδοτήσεις δεν υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν ότι το ελάχιστο θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί να σεβαστεί απόλυτα το αποτέλεσμα του Ρίο συν 20. Επίσης, ως ελάχιστο, τα, τις αρχές της δρόμης για την ε, τροφιμική ασφάλεια, να καταπολεμήσει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα. Αυτός είναι, αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες των τελευταίων ετών, ότι δεν καταφέραμε καν να μειώσουμε την κερδοσκοπία για τα τρόφιμα και πρέπει να βρούμε μακροπρόθεσμα μέτρα για να αποσυνδέσουμε την ξηρασία με τους λοιμούς. Διότι σήμερα βλέπουμε ότι σημειώνονται λοιμοί στο νότιο Σαχέλ και στο νότιο κάτω από το Σαχέλ Επίσης υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, η ενδυνάμωση του συντονισμού μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και ανθρωπιστικής τιάφτης. Άλλο τεράστιο θέμα, ο έλεγχος της αρπαγής γεών. Έχουμε αυτή τη στιγμή 10 εκατομμύρια εκτάρια που αγοράζονται κάθε χρόνο από διάφορους μεγάλες εταιρείες, χώρες και τα θύματα της αρπαγής αυτής είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες που χάνουν έτσι τις καλλιεργήσιμες γέες τους για τη δημιουργία παραδείγματος χάρη αγροκαυσίμων και δημιουργούν νέες συνθήκες ανέχειας διότι δεν τις προστατεύουν οι υπάρχουσες νομικές δομές. Υπάρχει μια συμφωνία που μόλις υπογράφηκε αλλά είναι εθελοντική για την πλαισίωση αυτή της εξέλιξη για τις ΓΕΕΣ και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και επίγον. Πρέπει επίσης να ενδυναμώσουμε το ρόλο της ΟΝΟΚΑ για το συντονισμό της, ανθρωπιστικής, της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και κυρίως, κατά προτεραιότητα μάλλον, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Ένωση στο κέρας της Αφρικής και να καταπολεμήσουμε τη ρίζα των σειράξεων που σημειώνονται εκεί, που είναι και θέμα τροφιμικής ασφαλείας. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο, να μην το λάβει. Α, θέλετε το λόγο, μάλιστα. Τότε έχετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, εγώ τα υπογραμμίζω απόλυτα, τα υποστηρίζω. Είχαμε την ευκαιρία πριν από ε, λίγες μέρες να συναντήσουμε την κυρία Helen Clark και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Μας είπε ότι πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μέχρι το 2015 καλύτερα τους στόχους χιλιετίες. όλα τα θέματα της ε, οικογένεια, του οικογενειακού σχεδιασμού είναι θέματα τα οποία τώρα αποκτούν μεγάλη σημασία και πρέπει να εργαστούμε για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά και με την κυρία Κλάρκ. Το πρόβλημα της κατάσχεσης των γεών στον τρίτο κόσμο μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Επιτροπή μας και να το αντιμετωπίσουμε με προτεραιότητα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Επιτροπή μας. Σίγουρα για την ομάδα μου θα πρέπει να είναι μία από τις ε, βασικές συνιστώσεις των στόχων της χιλιετίας στο θέμα της, ε, του οικογενειακού σχεδιασμού, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παράλληλα και το θέμα της κατάσχεσης γεών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, αν θέλει να θες. Α, η κυρία Στίφλερ προηγουμένως πάρα πολύ σύντομη κυρία Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Πρέντα που μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζολή για την ποιότητα της γνωμοδότησής της που αντανακλά πλήρω τη θέση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ο κύριος Πρέντα είναι ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ για τα θέματα αυτά. Στην, ε, για την ε, συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ λέει ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στα θέματα της ε, στρατηγικής της χιλιετίας και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σημείο δέλτα αυτής της γνωμοδότησης αναφέρεται στα συμπεράσματα του τέταρτου φόρουμ για την ε, βοήθεια επίτευξη των στόχων αυτών και επίσης για την ενίσχυση της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και τονίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη ε, τοπική λειτουργία των προγραμμάτων και ευθυγράμμιση με τις εθνικές στρατηγικές και μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, ε χορηγών για να έχουμε μικρότερο κόστος απόδοσης βοήθειας. Στην 68η λοιπόν Γενική Συνέλευση θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις του Φόρεμ του Μπούσεν, όπως αναφέρεται. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε μια χωριστή ψηφοφορία για το σημείο Β και μια χωριστή ψηφοφορία επίσης στο σημείο Ζ. Και σας τα λέω αυτά και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την επιστροφή της κυρίας Εύα Ζολή. Ήμουνα πάρα πολύ ε, κοντά της σε αυτή την εκστρατεία και ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολη η εκστρατεία η προεκλογική που έλαβε χώρα στη Γαλλία. Η Κομισιόν, η κυρία Φρανσούας Μωρό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ε, εισαγωγή για το σχέδιο αυτογνωμοδότησης. Η Κομισιόν αρχίζει να σκέφτεται τι θα γίνει μετά το 2015. Είναι σαφές όμως όπως φάνηκε και από πολλές παρεμβάσεις φουλευτών, για μας αυτό το οποίο προέχει είναι να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας όπως ισχύουν αυτή τη στιγμή μέχρι το 2015. Υπήρξαν πράγματι σημαντικές πρόοδοι, σίγουρα σε ορισμένε χώρε, σε ορισμένε περιοχέ του κόσμου τα πράγματα πήγανε πολύ καλά. Αλλού αυτό δεν ισχύει τόσο. Υπάρχουν κάποιοι δείκτε οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει. Αναφερθήκαμε στο θέμα της, ε, ε του οικογενειακού σχεδιασμού αλλά πρέπει να μην ξεχάσουμε και θέματα όπως η ένδυα, η καταπολέμηση της ένδυας, η αντιμετώπιση της πείνας που είναι σημαντικά θέματα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Δεύτερον, ακόμα και αν είχαν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι το 2015 για το στόχο υπαριθμών 1, δεν θα είχαμε παραπλώς μειώσει την ένδυα κατά το ίμιση. Η πρόκληση, επομένω παραμένει και επέκεινα του 2015 και είναι πάρα πολύ σημαντική. ως Επιτροπή, εμείς έχουμε σαν στόχο να προετοιμάσουμε μια ανακοίνωση για την αρχή του επόμενου έτους, η οποία βέβαια θα γίνει μετά από μια δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσουμε στις επόμενες εβδομάδες. Και εμείς παρακολουθούμε και τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά. Ο Γενικός Γραμματέας μας ζήτησε να προχωρήσουμε σε διαβουλεύσεις στις χώρες αυτές που είναι οι πιο φτωχές χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών και αναφέρατε και τη σημασία του να υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα ξεπεράσει αποκλειστικά και μόνο τους κρατικούς φορείς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μια αντιμετώπιση από τη δική μας πλευρά, όχι αναμονής, αλλά να ακούσουμε τις απόψεις όλων αυτών των φορέων. Αυτή είναι η σωστή πολιτική αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί να είναι διαφορετικό το πλαίσιο από το πλαίσιο που ίσχυε όταν έγιναν δεκτοί οι στόχοι της χιλιατίας πριν από 10 χρόνια, είναι στόχοι οι οποίοι έχουν διατυπωθεί ουσιαστικά από την ομάδα των χορηγών. Αυτή τη φορά όμως είναι απαραίτητο να έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι πιο συμμετοχική και πιο οικουμενική. Αυτό μας φαίνεται πολύ σημαντικό. Πέραν λοιπόν της ε, προετοιμασίας της θέσης της, η Κομισιόν θέλει να προσπαθήσει να συνενώσει τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από μια κοινή προσέγγιση, γύρω από κοινές αρχές, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση η ίδια δεν θα ξεκινήσει πριν από τον επόμενο χρόνο, κατά πώς φτάνοντα μέσα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, αλλά ούτως ή άλλως θα υπάρξουν ορισμένα μπλοκ διαπραγματεύσεων τα οποία θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αναφερθήκατε στην προετοιμασία της συνδιάσκεψης Ρίο 20 που θα αντιμετωπίσει πολλά θέματα που έχουν μεγάλη σχέση με μια παγκόσμια ατσέντα για, το 2000, για πέρα από το 2015. Η συνδιάσκεψη του Μπουσάν παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο τα αποτελέσματα του πάνελ υψηλού επίπεδου σε σχέση με την ενέργεια για όλους και αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά σαν σημεία αναφοράς τα οποία θα είναι και αυτά στοιχεία της συζήτησης για το 2015 και μετά. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα για το τι θα γίνει μετά το 2015, κάποια σημεία εμπλοκής μας ενδιαφέρει λοιπόν να μην έχουμε ε, προβλήματα εάν η συνδιάσκεψη για το Ρίο συν 20 χρόνια δεν επιτύχει τους στόχους τους. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις προτάσεις ε, τις, ε, να επιτευχθούν στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά όλα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν και με τη διαδικασία μετά το 2015. Η, εξωτερική, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θέλει να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κριστίνε Περόν, είμαι επικεφαλής της ε, μονάδος για τα πολυμερή θέματα αλλά παρακολουθώ και τα ζητήματα του ΟΗΕ, την προετοιμασία για την 67η Γενική Συνέλευση. Προφανώς υποστηρίζουμε ιδιαίτερα το έργο του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε συζήτηση με τον εισηγητή μέσα στα πλαίσια της ομάδας εργασίας. Έχουμε μόλις αρχίσει την επεξεργασία των προτεραιοτήτων, αλλά όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε είναι ζητήματα τα οποία θα λάβουμε υπόψη για τη διαδικασία του 2015 και θα τα συνδέσουμε με τα θέματα της ε, ε, διάσκεψης Ρίο συν 20 που περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, την ε, ε, ενέργεια, όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ε, αναπτυσσόμενο χώρο και φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την <clears throat> ανθρωπιστική πρόσβαση. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση και να είμαστε σε ένα σωστό διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε σήμερα. Η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει στις 31 Μαΐου. Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σημείο για τα χρηματοδοτικά μέσα. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό μηχανισμό για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά το κόσμο. Είναι έκθεση του κυρίου Φίλιπ Κάσμαρεκ. Δεν είναι εδώ. Τον αντικαθεστά όμως ο κύριος Λίσεκ. Παρακαλώ κύριε Λίσεκ, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Σύντομο παρακαλώ. Okay, this works. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι όντως πολύ σύντομος. Ο κύριος Κατσμάρικ, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να έρθει εδώ σήμερα. Οπότε, εγώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα σας παρουσιάσω την ε, πρότασή του για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού για την προαγωγή της ε, δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Είναι πρόταση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο εισηγητής ε, λέει ότι στην απόφαση πρέπει να φαίνεται η δικιά μας η δέσμευση προκειμένου να παλύψουμε τη φτώχεια και να προωθήσουμε μια προσέγγιση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αρχίσω παρουσιάζοντάς σας κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όπως γνωρίζετε, οι οργανώσεις αυτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία και στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Ο κύριος Κατσμάρακ υπογραμμίζει στην γνωμοδότησή του την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος τους μέσω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να παρατηρούν τις εκλογές και προκειμένου ε, το λέει στα άρθρα 1 και 2, να είναι παρατηρητές. Το άρθρο 2 λέει ότι υπάρχει μεγάλη πρόκληση ε, για τις ε, περιφερειακές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα για τις παρατηρήσεις. Όπως ξέρετε, 25% είναι ένα όριο για την παρατήρηση στις εκλογές. Αυτό ισχύει ήδη με την εφαρμογή του σημερινού DHR. Ο εισηγητής το λέει στο άρθρο του 2. Σημείο 3 τώρα, για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, δημοκρατική διακυβέρνηση. Είναι πάντα χρήσιμο να τονίζουμε περισσότερο αυτά τα θέματα. Πολλές φορές αναφέρονται και ιδίω στο άρθρο 2. Είναι η προσέγγιση δηλαδή βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης και η ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών. Υπάρχει και μία μνήα στην ανάπτυξη γιατί μόνο τότε μπορεί πραγματικά πλήρως να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γίνεται μια τέτοια μνήα και εδώ, πάλι στο άρθρο 2, για την πρόθεση της ανεξαρτησίας και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Τέλος, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική. Μου ζήτησε ο συγκητή να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ανησυχίες του όσον αφορά το θέμα αυτό. Υπάρχει κάποια περιθωριοποίηση. Πιστεύει ότι η αναπτυξιακή μας πολιτική βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη και για το PCD. Ευχαριστώ. Κυρία Κάισερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Θα αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία που προτείνει ο κύριος Κάτσμαρκ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά αναφέρονται στο κείμενό του. Ευχαριστώ τον κύριο Κασμαρέκ για την γνωμοδότησή του, πρώτα απ' όλα γιατί όντως παρουσιάζει πολύ καλά το νέο αυτό μέσο. Υπογραμμίζω όμως και υπογραμμίζω και εγώ ότι το μέσο αυτό υπογραμμίζω και ο Κάσμα, τον οποίο εκπροσωπώ δηλαδή εδώ, ότι περιλαμβάνει κάποιες δυσκολίες. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεισέφερε όλος ιδιαίτερος, ιδίως όταν βλέπουμε την, ε, ε, την Αραβική Άνοιξη, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να ανυψώσει την εικόνα της στις περιοχές αυτές. Το μέσο αυτό εξάλλου επικεντρώνεται περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις με τις οποίες ίσως δεν συμφωνούν οι κυβερνήσεις τους. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό μέσο το οποίο πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για να φέρει σε πέρα στο ρόλο του. Ο κύριος Κάσμαν επιμένει επίσης και σε κάτι άλλο. Λέει ότι η πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά πάντα της Αναπτυξιακής Επιτροπής, αλλά όχι μόνο, και άλλων πολιτικών, της εμπορικής για παράδειγμα, και ότι αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Όλες αυτές είναι θετικές πτυχές λοιπόν σε σχέση με αυτά που έχει πει ο κύριος Κάσμαρεκ και σε σχέση με αυτά τα οποία πρέπει να είναι το μέσο. Τώρα βέβαια εδώ δεν μιλάω ε, από αυτά που είπε ο Κάσμαν. Σας λέω κάτι επιπλέον, ότι προσοχή να μην αντικαταστήσουμε την πρωτοβουλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα με αυτό, αλλά να συμπληρώσουμε την πρωτοβουλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δρώντας πιο γρήγορα ή με άλλες πρωτοβουλίες πιο σύντομες. Έτσι κι και τα δύο χρειάζονται. Λέει ο κύριο Κάσμαν ότι υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών κτλ. Εδώ τώρα το ζήτημα του κύριου Κάσμαν που είναι πολύ σημαντικό είναι το 25% για αποστολή παρατηρητών στις εκλογές. Εγώ δεν έχω τα νούμερα βέβαια στο κεφάλι μου, αλλά θυμάμαι ότι όταν κάναμε μία έκθεση για παρατηρητές με τον κύριο Σαλαφράκα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τότε είχαμε βάλει κάποια οροφή. Είχαμε πει, εντάξει δεν είναι απόλυτα σταθερό, αλλά δεν θα πρέπει να είναι πάνω από δεν ξέρω αν ήταν 25% για αν αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με αυτό που λέμε στη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω όποιο αντικαθιστά εδώ τον κύριο Κασμαρή και ίσως να μπορεί να μου πει αυτό το 25% τι σημαίνει. Σημαίνει κάποια αύξηση σε σχέση με αυτό που είχαμε. Σημαίνει ότι κρατάμε το, τη σημερινή οροφή. Αν διατηρούμε τη σημερινή οροφή τότε μήπως προκαταλαμβάνουμε άλλου είδου βοήθεια που ήταν ε, βοήθεια στα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών κτλ. Να μου το απαντήσετε παρακαλώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει ο κύριος Κάσμαν ευχαριστεί ειλικρινά τον εισηγητή για την προσέγγιση του αυτή, η οποία διέπεται από συνοχή και είναι πολύ καλά κατανοητή. Τώρα εντάξει, εγώ βέβαια βγήκα κάπως από το κείμενο που μου είχε δώσει ο κύριος Κάσμαν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωραία, το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, λέει Πρόεδρο, ο κύριο Ρώσα, αντικαθιστά, ε, εκπροσωπή μάλλον Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατσουμάρεκ κλείπει βέβαια, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμπλησία απόψεων. Επίσης νομίζω ότι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί συμπληρώνουν το κείμενο χρήσιμα Όσο για τα σχόλια της κυρίας Ντεκάιζερ και τις τροπολογίες της, εξ ονόματος του κυρίου Κάσμαν, συμφωνούμε με αυτά που είπε. Γι' αυτό, παραδείγματο χάρη, στην τροπολογία 4 γίνεται λόγος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτό ακόμη και δεν είναι σωστό επομένως να βρίσκεται στο σκεπτικό ενός νομοθετήματος. για το ερώτημα του 25% αυτό είχε ήδη προβλεφθεί, προβλεπόταν στον προηγούμενο κανονισμό και απλώς παρέμεινε. Ο κύριος Κατσμάρεκ απλώς επανέλαβε την ίδια διατύπωση και συμφωνούμε και με αυτό. Βάζει ένα ανώτατο όριο, σωστό είναι αυτό, για τους στόχους που θέτει. Για το τα άλλα, τις άλλες τροπολογίες δηλαδή, συμφωνούμε σχεδόν με όλες και γι' αυτό μπορώ να πω ότι δεν έχουμε άλλα σχόλια σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρίσεκ για να καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι και θα τα διαβιβάσω στον κύριο Κατσμάρκ γιατί δεν είμαι εγώ αρμοδιότερος να μιλήσω εκ μέρους του. Εκείνος έχει συντάξει το κείμενο και δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο, θα του μεταβιβάσω όλα αυτά που ακούστηκαν. Σας υπενθυμίζω, όχι, ότι η διάθεση στι στις 13 Μαΐου, στις 30 Μαΐου λίγη η διορία κατάσταση των και θα ψηφίσουμε στις 4 Ιουνίου ενώ η ΕΠΕΞ θα ψηφίσει στις 10 Ιουλίου. Τώρα πάμε στις ψυχοφθορίες. Παρακαλώ να, φέρετε, να βγάλετε τις κάρτες σας από τα πορτοφόλια. Ευχαριστώ. Ένα τεστ να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες σας. Le Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Όχι. Εντάξει, συνεχίζει να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 18 ψήφισαν, 14 υπέρ, 3 κατά μία αποχή. Εντάξει. Madame comment D'accord. Madame Costello, vous avez quelque chose à nous dire Κυρία Κοστέλο, θέλετε να πείτε κάτι? Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Κοστέλο. Έχω πρόβλημα με την κάρτα μου. Να προσπαθήσουμε και πάλι Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν και πάλι. Madame Costa. Ça marche. Ça marche C'est un votant de plus. C'est bon Εντάξει. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Τροπολογία 19 με χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F, σίγμα τα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, 22, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. «25». Θέλετε έλεγχο στην 24, βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία για την 24. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται όμως. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικά στην ε, γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα δεκτή. και συγχαρητήρια στην κυρία Λετβίν που είναι γνωστή για την τις προσπάθειές της για τη βιώσιμη αλία. Τώρα θα ψηφίσουμε την συμπερίληψη των υπερποντίων χωρών και εδαφών. Είναι η έκθεση του κ. Πόγκα, δεν έχει τροπολογίες. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την ε, έκθεση αυτή. Ψήφισατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, μία ψήφος κατά. Γίνεται δεκτή η έκθεση. Συγχαρητήρια στον κύριο Πόγκα. Ψηφίζουμε τώρα τη δική μου έκθεση σε σχέση <clears throat> με την σύσταση του Κοινοβουλίου για την 67ο Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, δεύτερη τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για την έκθεση σας σύνολο, άρχεται ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Ομόφωνα δεκτή. Ωραία. Τελειώσαν οι ψηφοφορίες. Τοποθετήστε στο πορτοφόλι τις κάρτες σας. Εξετάζουμε τώρα την εντολή για τον τριγωνικό διαλόγου στις 23 ε, Μαρτίου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό του 2013 παρουσία του κυρίου Λαβιά του Γενικού Εισηγητή για τον προϋπολογισμό 2013. Τώρα η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει το σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2013. Ο κύριος Λαβιά έχει δημοσιεύσει το σχέδιο έκθεσή του για την εντολή του Κοινοβουλίου για τον τριγωνικό διάλογο, πρέπει να προετοιμάσουμε και τη γνώμη της Επιτροπής μας απαντώντας σε αυτό το έγγραφο. Παρακαλώ τον κύριο Γκέι Μίτσελ, που είναι ο εισηγητής μας, να μας παρουσιάσει τις γενικές γραμμές της γνωμοδότησής του. Έχετε το λόγο κύριε Μίτσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω εδώ εκ νέου στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή μας. για τον προπολογισμό. Κάναμε μια πρώτη συνάντηση των εισηγητών την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λαβία για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνεννόηση και για την παρουσία του και σήμερα. Έχει κάνει πολλά για αυτή την έκθεση. Προσπάθησε να ακούσει όλα όσα του συνέστησαν. Την περασμένη εβδομάδα είπα ότι δεν μου αρέσουν οι περικοπές στο DCI. Ξέρω ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι κατά 1,3% υπάρχει αύξηση των κοντιλίων του DCI και, αλλά οι περικοπές συνδέονται πιο συγκεκριμένα με την υποχρησιμοποίηση των κοντιλίων για συγκεκριμένα σχέδια. Ως προς τις αρνητικές προτεραιότητες μπορεί να συμφωνούσαμε για περικοπές σε ορισμένους τομείς, όπως την Ιεμένη, το Ιράκ και το Ιράν, όπου υπάρχουν προβλήματα απορρόφησης ορισμένων προγραμμάτων, αλλά για άλλες θέσεις όπως την Ασία, την Κεντρική Ασία Νομίζω ότι οι περικοπές γίνονται χωρίς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή αιτιολόγηση. Ίσως λοιπόν η Κομισιόν εδώ να μπορεί να μας δώσει ορισμένες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες γιατί περικόπτονται τα κονδύλια της Ασίας και της Κεντρικής Ασίας. Επίσης θα μπορούσε να μας αποσαφηνίσει αν η αύξηση των θεματικών προγραμμάτων του DCI για το περιβάλλον και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι πράγματι προσθετική, πρόσθετη χρηματοδότηση. Γιατί η χρηματοδότηση τομέων κλειδιών όπως η παιδεία δεν θα έπρεπε να συγχέεται με την κλιματολογική αντιμετώπιση. Φυσικά και αυτή τη θέλουμε, αλλά όχι εις βάρος της υγείας και της παιδείας. Με ανησυχούν ιδιαίτερα και οι περικοπές για τα διοικητικά έξοδα για την τεχνική βοήθεια. Είδα τις ποσοστώσεις και ξέρω ότι στην εποχή που ζούμε πρέπει να είμαστε λογικοί ως προς τον τρόπο χρήσης των πόρων που διαθέτουμε, αλλά οι δραστηριότητες αυτές χρειάζονται και για αξιολόγηση και για άλλους σκοπούς στο DCI 2 δεν ξέρουμε ακόμη αν όντως δαπανίσαμε το 20% για τα βασικά προγράμματα υγείας και παιδείας. Χρειάζονται λοιπόν πλήρη κριτήρια αξιολόγησης που χρειάζονται και για την Ένωση, για τις αρχές του προϋπολογισμού Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και γενικότερα είναι χρήσιμο και για τους πολίτες. Ιδιαίτερα ξέρω ότι οι υπάλληλοι του DCI στον προπολογισμό του 2013 είναι κάτι που με ανησυχεί. Το 11 η Κομισιόν ζήτησε 18 πρόσθετα πλήρη μέλη για να διασφαλίσει, λέει, τη σωστότερη διαχείριση πολλών προγραμμάτων μικρής εμβέλειας. Δηλαδή, για να υπάρξει καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση για να ξέρουμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται και για να υπάρχει, καλύτεροι λογαριασμοί. Αυτό ήταν από το σχέδιο προϋπολογισμού του 12. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν. Γιατί μετά περιέκοψε κατά 51 τον αριθμό αυτών των υπαλλήλων. Αφού αυτοί είναι οι λόγοι για την αύξηση το 12, γιατί ποιοι είναι οι λόγοι για την περικοπή. Εγώ δέχομαι τη διατήρηση των επιπέδων για την ανθρωπιστική βοήθεια και την κατεπίγουσα βοήθεια, για το αποθεματικό δηλαδή, γιατί πρέπει η Ένωση να μπορεί να κινητοποιήσει χρήματα σε ανταπόκριση τυχών διεθνών ανθρωπιστικών κρίσεων που συνεχώς και αυξάνονται και πολλές φορές απρόβλεπτα. Τέλος, Πρόεδρε, ο κατάλογος για την κατάσταση των προγειών λύγει την Τετάρτη. Εγώ θέλω να καταθέσω πολλές για τομείς που νομίζω ότι δεν έχουν ακόμη λυθεί τα πράγματα και θα ήθελα η διορία να παραταθεί αν νομίζουν ότι θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κορτές Λαστρά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι ο προϋπολογισμός 2013 πρέπει να τα αποκρίνεται στον κύριο στόχο που είναι η μείωση της ένδυας. Και αυτό με φόρο ανάπτυξη, άρα ακριβώς η οικονομική ανάπτυξη είναι το βασικό στοιχείο. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια συνδέεται πάρα πολύ με την εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζομαι να είναι φιλόδοξος. Συμφωνούμε με τον ειδικό εισηγητή όσον αφορά τους ε, στόχους της, που θέλει για τις υποχρεώσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε δαπάνες κάτω από το προβλεπόμενο όριο και ότι το DCI όσον αφορά τις πληρωμές είναι χαμηλότερο από ό,τι για το 2012. Πιστεύουμε επίσης ότι οι πόροι που πάνε στην ανάπτυξη πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μείωση της ένδειας στην βελτίωση των συνθηκών ζωής. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε σε συνεργασία με άλλους δόρυτες για να είμαστε ακριβώς αποτελεσματικοί. Ε, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για άλλα προγράμματα πιο μικρά, σε συνεργασία με τους κύριους φορείς, όχι απαραίτητα κρατητούς, με τον ιδιωτικό τομέα με τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους τοπικούς συνεταιρισμούς, για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει επίσης περισσότερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων και συνοχή με μηχανισμούς που να στοχεύουν και τις κλιματικές αλλαγές της υπονάπτυξη χώρες. Επίσης, με ικανοποίηση βλέπουμε και την πρόταση για αύξηση των επενδύσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού που έχει να κάνει με ε, τα άτομα και πιστεύουμε ότι το σημείο αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι πολύ σημαντικό και οι προηγούμενες υποχρώσεις από το, για το DCI οι πόροι του πρέπει να πηγαίνουν στην υγεία και τη βασική εκπαίδευση με ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας που ακόμα δεν έχουμε πετύχει, κάθε άλλο. Και τελειώνω με το εξή. Ευρωπαϊκή συνένεση για την ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να είναι το στοιχείο προς το οποίο προσανατολιζόμαστε. Με βασικά στοιχεία την υγεία και την εκπαίδευση. Και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό μέσο ώστε να πετύχουμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη με τη στήριξη μάλιστα της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων εγκαρσίων σημαντικών θεμάτων όπως είναι η ισότητα των δύο φύλων. Και η αντιμετώπιση του AIDS. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Δεν ξέρω ποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κάρλο Χέι. Έχω εδώ. Η κυρία Γιάννα Μπλάτισλαβ. ή ο κύριος Πάρτβας. Μην πέσετε κιόλα, μην πέσετε κιόλα, γιατί σκόνταψε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Συγγνώμη πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο προπολογισμό του 2013 διαδικαστικό λέει ο κύριο Μίτσορ. Σα είπα ο συνάδελφο ποια θέματα έθιξα προηγούμενα στην παρέμβασή μου. βεβαίω. Ελπίζω ότι τα έχω πάρει όλα αυτά που είπατε. Ο προπολογισμό του 2013 είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός του τωρινού πολιετούς πλαισίου και επίσης είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητος όπως σε όλα τα κράτη-μέλη μας και εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό ο οποίος θα περιορίσει τις πιστώσεις πληρωμών. Για να κρατήσουμε λοιπόν όχι μόνο το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, αλλά και τις προτεραιότητες που είχαμε θεσπίσει για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, όπου αυξήσαμε τη χρηματοδότηση κατά 45,9 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Επίσης, σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονίας, ιδίως στη Νότια Μεσόγειο, έχουμε εφαρμόσει αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο, προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την Αραβική Άνοιξη. Χρειάστηκε λοιπόν να περιοριστούμε σε ορισμένα προγράμματα και για να το επιτύχουμε αυτό ακολουθήσαμε μια μέθοδο η οποία βασίζεται ουσιαστικά στο επίπεδο απορρόφησης των κονδυλίων. Εξετάσαμε λοιπόν όλα τα προγράμματα, ιδίως τα προγράμματα που έχουν υπόλοιπα προς απορρόφηση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί, είτε γιατί είναι πολλά ακόμα έργα τα οποία δεν έχουν συναυθεί απαραίτητε συμβάσεις ή γιατί είχαν γίνει συμβάσει αλλά δεν είχαν γίνει καταβολές των πληρωμών. Βλέπουμε ότι ορισμένα προγράμματα, ιδίω στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, είχαν προβλήματα απορρόφησης είτε και πάλι όπως λέω διότι δεν ενδιαφερόντουσαν τα ε, κράτη της Ασίας και για τα προγράμματα αυτά είτε γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους. Μέσα στον προϋπολογισμό αυτό λοιπόν έχουμε υπολογίσει όσο μπορούσαμε καλύτερα τις πιστώσεις πληρωμών για να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε θα τηρήσουμε όλες τις δεσμεύσεις μας που είναι ήδη νομικά ισχυρές αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε πλεονάσματα. Θα υπάρξουν και προσαρμογές που θα γίνουν του χρόνου επί τη βάση των πραγματικών αναγκών. Αλλά θα παρεύουμε και μεταφορές πιστώσεων αν αυτό είναι απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη γραμμή Ασία-Κεντρική Αμερική, έχουμε προβλήματα απορρόφησης. και μετά από την ανακοίνωση Agenda for Change θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά τα προβλήματα. Για τους λογιστικούς ελέγχους και την ε, αξιολόγηση, εδώ, είμαστε έχουμε για τις περισσότερα, τα περισσότερα προγράμματα συμπερίληψη αυτών των γραμμών μέσα στο πρόγραμμα και όχι σε χωριστή γραμμή του προπολογισμού. Και έτσι οι χρηματοδοτήσεις αυτές πηγαίνουν στα λειτουργικά κονδύλια και δεν υπάρχει χωριστή γραμμή στον προπολογισμό. Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Σα Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος. Περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα για να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κυρία Μίτσελ, ναι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ένα τεχνικό πρόβλημα υπάρχει εδώ. Εάν δεν έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες μέχρι το μεσημέρι της 16ης του μηνό, ε, δεν θα μπορούν να μεταφραστούν. Είχα πει μεσημέρι της 17 η Μαου, ελπίζω θα συμφωνήσετε να είναι 16 το μεσημέρι για να προλάβουν να μεταφραστούν. Καταλαβαίνω όλα αυτά που είπε η Κομισιόν, καταλαβαίνω την ανάγκη να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη χρήση των πόρων μας σε συνθήκες όπω οι σημερινε, Αλλά επειδή είμαστε σε αυτήν την κατάσταση αρκετά χρόνια, δεν καταλαβαίνω γιατί το 2012 η Κομισιόν ζήτησε πρόσθετο προσωπικό για να εξασφαλίσει την καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση μικρών χορηγιών βάσει του προγράμματος για την ε, ανάπτυξη και μετά έχει περικόψει για το 2013 τον αριθμό του, των μελών του προσωπικού κατά 51 άτομα. Δεν θα έχουμε λοιπόν σωστή δημοσιονομική διαχείριση και λογοδοσία Πώς λοιπόν τα συμβιβάζετε όλα αυτά. Γιατί τα μέτρα λιτότητας που έχετε εφαρμόσει είναι πράγματα τα οποία ξέρετε ότι θα εργαστείτε να τα κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οριακή ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών 17 Μαΐου λέει η Πρόεδρος. Ναι, ναι, δεν κατάλαβα και καλά. Νομίζω ότι είχαμε γλιτώσει μια μέρα. Όχι, είναι 16 Μαΐου, πράγματι. 16 Μαΐου το μεσημέρι. Ο κύριος ε, Μιτσέλ έδεσε ένα σαφές ερώτημα προς την Κομισιόν. Θα ήθελε να ξέρει τι νόημα έχει να φτιάξετε 17 θέσεις για το DCI. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Euh, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρόκειται για 17 θέσεις που δημιουργήθηκαν πριν από τρία χρόνια για το Food Facility. Τελείωσε όμως αυτό. Επρόκειτο για θέσεις προσωρινές, για τρία χρόνια μόνο. Οι θέσεις αυτές δεν υπάρχουν συνεπώς πια. Αποτελεσματικά. Συνεπώς, όλες οι αντιπροσωπείες που υποφελήθηκαν Τώρα πια δεν έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις θέσεις. Ήταν ε, προσωρινού χαρακτήρα, προσωρινής διάρκειας θέσεις. Κύριε Μίτσελ, μα συγγνώμη, εγώ δεν συμφωνώ, ήμουν εισηγητής για τον κανονισμό αυτό και για τον DCI και το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 18 επιπλέον και για το 2012 είπε προκειμένου να υπάρξει χρηστή η οικονομική διαχείριση για τον DCI. Αυτά λέει το σχέδιο προπολογισμού για το 2012. Συνεπώς, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μήπως θέλετε να μας απαντήσετε, έχετε στοιχεία για να μας απαντήσετε, να δώσετε απάντηση στις διευκρινήσεις. Ε, πρόκειται για θέσεις για την διαχείριση πολλών προγραμμάτων ε, που καλύπτονταν από μικρά ποσά. Αν δεν είσαστε σε θέση τώρα να μας απαντήσετε, μπορείτε ίσως γραπτά να το κάνετε, να θέτω χρόνο στη γραμματεία. Εκπρόσωπος Επιτροπή. Ναι, προτιμώ να απαντήσω γραπτά, γιατί ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιες θέσει. μιλάει ο κύριο Μίτσελ. Ωραία. Συμφωνούμε τότε. Αυτό θα κάνουμε. Καλώς. Συνεπώ, τελείωσε αυτό το σημείο. Και έτσι περνάμε τώρα... Ο κύριος Σόρενσεν, καλώς θα ήταν, καλό θα ήταν να έρθει εδώ. Ελάτε παρακαλώ κύριε Σόρενσεν να καθίσετε δίπλα μου. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τις επικαιρότητε. Έχουμε μαζί μας τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Πρόκειται για την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία και την κατάσταση των Συρίων προσφύγων στην περιοχή. Φυσικά και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ όλους μας στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής. Ο Ασάντ Ελμπασάρ, όπως γνωρίζουμε όλοι, σκοτώνει τον κόσμο του. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι τύχη επιθυλάσετε σε όλους αυτούς τους Σύριους πρόσφυγες οι οποίοι πάνε στην Τουρκία ως επιτοπλίστων αλλά και στην Ιορδανία και ακόμα και στο Ιράκ. Συνεπώς, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω εδώ τον κύριο Σέρενσον, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή. Και εγώ θέλω να ξέρω κατά πόσο η ανθρωπιστική μας βοήθεια χρησιμοποιείται καλά. Τι προβλέπετε για να βοηθήσουμε αυτούς τους μάρτυρες της συλλογική μας ανικανότητας. Ευχαριστώ πολύ. Τα μάλα σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που επανήλθατε και είσαστε ενεργοί εδώ και όχι εκεί. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι στην Επιτροπή αυτή. Θέσατε τον δάκτυλόν σας επί των τύπων των ύλων αναφερόμενοι σε κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Αποτροπιαζόμαστε, γιατί οι τελευταίες εκθέσεις από τη Συρία δεν μας δίνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξία. Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι είναι μία εξέλιξη η οποία διολυσταίνει σε μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Δεν ξέρω τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι αυτή την κατάσταση σίγουρα δεν πάει προς την καλή κατεύθυνση. Έχουμε μία σύγκρουση που έχει αντιμέτωπους πάρα πολλούς, πάρα πολλές ομάδες του πληθυσμού και υπάρχουν πεπειραμένοι παρατηρητές που γνωρίζουν καλά τη Συρία και έχουν ζήσει εκεί, μας λένε ότι όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία είναι σχεδόν μη αντιστρεπτή. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψει αυτή την πορεία που θα οδηγήσει σε μια κατάσταση παραδεταμένης κρίσης και σύγκρουσης. Ως υπεύθυνο για τα ανθρωπιστικά θέματα, εγώ κρατάω μια θέση μεσοβέζικη. Γιατί ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε ως τον ατόν πιο ουδέτεροι, όχι επειδή μας αρέσει αυτό που βλέπουμε, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε ουδέτεροι ως μια ανθρωπιστική αρχή. Πρέπει να μείνουμε ανεξάρτητοι και ουδέτεροι, γιατί η δράση μας απαιτεί αυτή την ουδετερότητα και την αμεροληψία για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση επιτόπου. Δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και ανησυχία όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στον πολιτικό στίβο. Προσπαθούμε όμως συγχρόνως να πείσουμε τις διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές ότι εμείς ως η ανθρωπιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια ειδική ε, αποστολή. Δεν είναι το βασικό θέμα το αν είμαστε μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακολουθούμε την οδό της ουδετερότητας. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια αξιολόγηση αναγκών και να έχουμε πρόσβαση στον πληθυσμό. Να μην φοβόσαστε ότι έχουμε διαφορετική ατζέντα. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για να το κάνει κανείς πραγματικότητα. Υπάρχουν καχυποψίες, κάθε είδου. Εγώ πολλές φορές έχω χρειαστεί να καταπιώ αυτά τα οποία θέλω, θα έπρεπε να πω σαν προσωπική μου γνώμη και να εξοραίζω τις δηλώσεις μου. Το κάνω αυτό όταν μιλάω <clears throat> στον ε, πρεσβευτή της Συρίας στη Γενέβη δίνω έμφαση στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία και κάνω μια έκκληση σε αυτούς και μου λένε εσείς οι ανθρωπιστές έρχεστε εδώ γιατί θέλετε να πετύχετε κάτι άλλο. Πώς θα εμπιστευτούμε ότι δεν θα παρέμβετε σε αυτή την κατάσταση. Είναι λοιπόν ένα πολύ πολύπλοκο σενάριο. Αρκετά νωρίς μετά από τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο, αλλά και επειδή θεωρούσαμε ότι τα πράγματα δεν προχώρησαν αρκετά γρήγορα στο επίπεδο το ανθρωπιστικό, και θα σα εξηγήσω και γιατί δεν γινόταν αυτό, εμείς θεωρήσαμε ότι μια κάπως διαφορετική στάση υπήρχε από ορισμένου χορηγούς, οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί, γιατί ήδη μέσα στη Συρία για πάρα πολύ καιρό, επειδή η Συρία έχει υπερήφανες ε, παραδόσεις του να υποδέχεται πρόσφυγες από το Ιράκ ή από την Παλαιστίνη, η χώρα αυτή έχει ένα μεγάλο πληθυσμό προσφύγων ήδη. 200.000 πρόσφυγες από το Ιράκ που τις, τους ε, καλύπτει η, η πάτη αρμοστία για τους πρόσφυγες Έχουμε περίπου μισό εκατομμύριο Παλαιστινίων που ζουν κοντά ή γύρω στη Δαμασκό και τους υποστηρίζει η ούρα. Και όλα αυτά τα άτομα έπρεπε να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε σε συζητήσεις με τους Σύριους, οποιαδήποτε άσκηση πίεσης, οποιαδήποτε προσπάθεια πειθούς για να κάνουμε κάτι για τον λαό τους, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που ε, ενέχει για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη Συρία. Υπάρχει λοιπόν αυτό ο κίνδυνο για τα ανθρωπιστικά θέματα. Ο τρόπο με τον οποίο προσπαθήσαμε να λύσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα ήταν να πούμε και στην ε, διάσκεψη Ισλαμικών κρατών και τον Αραβικό Σύνδεσμο ότι πρέπει να υπάρξει ένα τρόπο να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση τη Συρίας Πρέπει να γίνει δημόσιο ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανθρωπιστικό διάβλο μαζί με τον πολιτικό διάβλο. Χωρίς όμως να τα αναμίξουμε ιδιαίτερα τα δύο θέματα αυτά. Και εκεί είχαμε υποστήριξη από πολλούς εμπλεκόμενους για να φτιάξουμε το ανθρωπιστικό φόρουμ για την Συρία. <clears throat> που για δεύτερη φορά συνεδρίασε στη Γενέβη πριν από τρεις εβδομάδες. Το, ποτήρι βέβαια είναι για ορισμένου μισογεμάτο, για ορισμένου μισοάδιο. Δεν είναι μια εντυπωσιακή επιτυχία. Τις δύο φορές όμως που συνεδριάσαμε, δημιουργήθηκε μια κίνηση, μια ορμή που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο ανθρωπιστικό αυτό μέτωπο. Η πρώτη συνάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί οι φίλοι μας από τη Συρία δεν θέλαν ιδιαίτερα να συμμετάσχουν. Μετά από κάποια διπλωματία διαδρόμων ήρθαν τελικά να συζητήσουν μαζί μας και τα καλά νέα ήταν ότι 24 ώρες προηγουμένως ο Βάλεο είχε καταφέρει να πάει στη Δαμασκό και να έχει πρόσβαση εκεί. Θυμάστε τις ε, φωτογραφίες από το Χόμς και την Τέρα και εκεί που είχαν βομβαρδιστεί από το στρατό της Συρίας. Ήταν μια πρώτη ευκαιρία για, τους, ε, για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πέραν της Ερυθράς Μισελίνου που είναι εθνική οργάνωση της Συρίας και της ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και φυσικά και τον Ερυθρό Σταυρό που είχε μεγάλη δυσκολία πρόσβασης. Το γεγονός ότι ο Βαλωριέμος μπόρεσε να έχει μια πρόσβαση ήταν πολύ σημαντικό. Εμείς δεν θα συμμετείχαμε κανονικά σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά δεχτήκαμε να συμπροεδρεύσουμε μαζί με την Οργάνωση Ισλαμικών Κρατών και τον Αραβικό Σύνδεσμο για να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους φορείς του ΟΗΕ να μην είναι μόνοι. Η δεύτερη συνάντηση πριν από τρεις εβδομάδες επέτρεψε μία αποστολή εκτίμησης των αναγκών να ξεκινήσει. Γιατί αν πάτε στη Συρία και δεν ξέρετε πού χρειάζονται βοήθεια τα άτομα, ποιες είναι οι ανάγκες τους, πόσα νοσοκομεία έχουν ισοπεδωθεί, τι γίνεται σε διάφορα μέρη, κινδυνεύετε να παροχετεύσετε τη βοήθειά σας σε μέρη που υπάρχει λιγότερη βοήθεια και κυρίως κινδυνεύετε να θεωρηθείτε ότι είστε τμήμα της σύγκρουσης, ότι έχετε πάρει κάποια πλευρά. Και από εκεί τέρμα η ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ καλή ανάλυση εκ των προτέρων και πάλι το ποτήρι είναι μισοάδιο αλλά και μισογεμάτο. Μας αφήσαμε να πάμε εκεί και οι παρατηρητές μας μπόρεσαν να δουν και κάποιους αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης και να προχωρήσουν σε μια ανάλυση η οποία μπόρεσε να συζητηθεί. Ζητήσαμε την υπογραφή της κυβέρνησης της Συρίας και στο δεύτερο ανθρωπιστικό φόρουμ το μήνυμα ήρθε ναι, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα έκτακτο ανθρωπιστικό πρόβλημα, περίπου ένα εκατομμύριο άτομα τα οποία έχουν φύγει από τις αιστείες τους. Η πρώτη φορά που το αναγνωρίσαμε. Και πάλι αυτό δεν αποτελεί λύση. Πρέπει να δώσουμε συνέχεια και να έχουμε την κατάλληλη πρόσβαση και πάλι δεν είναι θέμα χρημάτων. Έχουμε με τη βοήθειά σας εκταμιεύσει 3 εκατομμύρια και μετά 7 εκατομμύρια και άλλα 10 εκατομμύρια. Όταν έχουμε καλύτερη πρόσβαση θα είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε σε εσά για να χρησιμοποιήσουμε το απόθεμα, το αποθεματικό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά όλα αυτά έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ότι μπορούμε να φέρουμε τα εφόδια που χρειάζεται σε διάφορα τμήματα της Συρίας. Όλα αυτά είναι λοιπόν αρκετά ταπεινά. Κάτι το οποίο είναι θετικό από αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτός ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της υπάτης αρμοστίας για τους πρόσφυγες στη Δαμασκό και ήταν υπουργό στην Τίνιδα μετά από την Αραβική Άνοιξη και είναι εμπειρογνώμων για τα θέματα της ε, Συρίας. Εγώ ξέρω κάτι, αλλά αυτός ξέρει πολλά περισσότερα. Και μας είπε, μην σπρώξετε πολύ τα πράγματα, χρειάζεται χρόνος, θα προσπαθήσω να μιλήσω με, τη, με, την, με τις Συριακές αρχές και τελικά καταφέρνει να υπάρχει κάποια μικρή πρόοδος ώστε η πάτη αρμοστήρια για τους πρόσφυγες και κάποια άλλοι χορηγοί μπορούν να ανοίξουν περιφερειακά γραφεία, στην ε, Χόμς, ε, στην Τέρα, στο Ιμπίλ και άλλα μέρη. Όχι ότι τώρα αυτά τα πράγματα μας δίνουν πολύ ελπίδα γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αλλά βλέπω ότι, ότι αυτές οι προσπάθειες αυτές, προσπάθειες ουδετερότητας αλλά παρόλα αυτά πίεση στην κυβέρνηση της Συρίας έχουν αποφέρει κάποιους καρπούς. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Και αν κάποιος έχει το μαγικό ραβδί και να πει εντάξει θα πάμε, θα προχωρήσουμε από τους διαδρόμους, θα φτιάξουμε buffer zones. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Η πραγματικότητα όμως είναι, και νομίζω ότι πρέπει να το δεχτούμε αυτό, η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Για μένα λοιπόν αυτό είναι το σήμα που με κάνει να πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθούμε με μεγάλη ισορροπία, να παρατηρούμε καλά τι συμβαίνει, να πιέζουμε, χωρίς όμως να μπούμε και στην παγίδα να προσπαθούμε να κάνουμε εμεί πολιτική μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί τότε η κυβέρνηση η οποία ελέγχει τις μεταφορές, την διανομή, θα κλείσει την πόρτα και θα την κλείσω όχι μόνο σε εμά, αλλά και σε άλλους παράγοντες εκεί. Ευχαριστώ τώρα να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε για να σας ενημερώσω καλύτερα. Πάντως να ξέρετε ότι όλα αυτά μας κάνουν να ξαγρυπνούμε τις νύχτες γιατί τα παρακολουθούμε. Είμαστε συνέχεια σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μας με όλους τους παράγοντες και προσπαθούμε να πάρουμε αυτό το στενό δρόμο που είναι ανάμεσα στην πολιτική και στην βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε κάτι, εσείς μιλήσατε πριν για τους πρόσφυγες, τους Σύριους, ε, και αυτούς τους φροντίζουμε στην Ιορδανία, στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε τα σύνορα Πηγαίνω στην Ιορδανία, στο Λίβανο και έχουμε κάνει και προσφορές στην τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να τους υποδεχθούν. Πρέπει να συγχαρώ αυτές τις γείτονες χώρες γιατί έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν τα δικά τους προβλήματα. Έχουν πολλά προβλήματα. Είναι και αυτή η υποπίεση. Αλλά εμείς είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε φυσικά και συμμετέχουν και αυτοί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Κάτι τελευταίο. Αντίθετα από τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου ξέρετε πό τι θέσεις έχουν τα διάφορα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η δικιά μου εμπειρία είναι ότι οι συνομιλίες με τους Κινέζους, με τους Ρώσους ήταν χρήσιμες δεν θέλουν να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Έχουμε πετύχει να μην έχει επιδεινωθεί περισσότερο η κατάσταση. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι τόσο οι Κινέζοι όσο και οι Ρώσοι, ιδιαίτερα οι Ρώσοι, ανθρωπιστικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να περάσει το μήνυμα σύμφωνα με την ανθρωπιστική ατζέντα που έχουμε. Αυτά έχω να σας πω κάπως σύντομα και από εκεί και πέρα ό,τι ερωτήσεις έχετε είμαι στη διάθεσή σας. Σας κατευχαριστώ. Κυρία Κάιζερ, Κάιζερ. Ευχαριστώ κύριέ μου για τις προσπάθειες που κάνετε. Προσωπικά πιστεύω ότι η στρατηγική σας διαχωρισμού του ανθρωπιστικού από το πολιτικό είναι ο μόνος δυνατός δρόμος. Είναι μονόδρομος που λέμε. Είναι βέβαια μακρύς ο δρόμος προς τον εκδημοκρατισμό και χρειάζεται αντοχή. Οποιαδήποτε άλλη λύση, απλούστερη ή γρηγορότερη, θα οδηγούσε σε περιφερειακή καταστροφή. Κατάλαβα καλά ότι σήμερα και στο εσωτερικό της Συρίας ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια έγιναν μερικά θετικά βήματα και είπατε ότι οι δωρητές και δωρήτριες μπορούν να ανοίξουν γραφεία αποκεντρωμένα στο Χόμς ας πούμε στην Τέρα και αλλού. Αυτό το επιβεβαιώνεται και τι φύσης είναι αυτή η βοήθεια γιατί μιλήσατε για κέντρα διανομής κλπ. Είναι ιατρική, είναι χρήματα σε μετρητά γιατί χρειάζονται και μετρητά. Τι είδους βοήθεια είναι, τι φύση είναι, θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Δεύτερον, κάνατε πολλές προσπάθειες για να πλησιάσετε την κυβέρνηση της Συρίας και για να την πείσετε για τη σημασία που έχει η αποστολή σας. Οι άλλες χώρες τι κάνουν γιατί τελευταία πήγαμε την κυρία Γκόμε στο Λίβανο όπου υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία ιδιαίτερα από το Χόμς γιατί είναι κοντά στα σύνορα η κυβέρνηση Μικάτη είχε καταγράψει περίπου 10.000 πρόσφυγες στα σύνορα στο βορρά, αλλά δεν είχε καταγράψει, ούτε θέλει να το πράξει, ούτε θέλει να βοηθήσει και να επιτρέψει στην Επιτροπή High Committee Relief άλλους τόσους που βρίσκονται στην ΠΚΑ. Στο Λίβανο λοιπόν, όπου υπάρχει κυβέρνηση που είναι υπέρ του Μπάσαρ και τουλάχιστον το Χεσμπολά την υποστηρίζει εκεί η ροή αυτή των προσφύγων είναι και ανθρωπιστικό θέμα αλλά και πολιτικό. Τις δύο τελευταίες μέρες έγιναν οι πρώτες ταραχές και θάνατοι προς την Τρίπολη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κατορθώσουμε, να χορηγήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και να διευκολύνουμε τις οικογένειες των προσφύγων για να μην υπάρξει και νέα ανάφλεξη. Πώς το βλέπετε λοιπόν ως προς την κυβέρνηση με κάτι. Γιατί όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργό του Λιβάνου, κύριος Μιχάτη μας εξέφρασε και την άποψη του Προέδρου Σουλεϊμάν εδώ στο Κοινοβούλιο. Και τον ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε και μας είπε δεν υπάρχει πρόβλημα, εμείς τα ελέγχουμε όλα. Δεν έχουμε κανέναν στην ΠΑΚΑ. Και αυτό είναι φυσικά δεν είναι σωστό. Δεν είναι αλήθεια. Τι μπορέσατε εσείς να κάνετε λοιπόν και πώς ακριβώς έχει το πρόβλημα και αλλού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιμποφάκελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε και σλοβενική διερμηνία, οπότε θα χρησιμοποιήσω την ε, μητρική μου γλώσσα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε πάλι μαζί μας, κυρία Σόλη. Ήταν παρόλα αυτά πάρα σημαντικός ο, ο ρόλος σας και παίξατε και σημαντικό ρόλο εκπροσωπώντας με κάποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Ντεκέιζερ. Είναι πολύ καλό το ότι μπορέσετε να κρατήσετε μια απόσταση από την πολιτική. Ίσως όμως είναι υπερβολική αυτή η απόφαση από την ε, ε, από την πολιτική της Συρίας ως Ευρωπαίοι βουλευτές και ως Ευρωπαίοι πολιτικοί θεωρώ ότι παραμένουμε σε ένα επιδερμικό επίπεδο. Έχουμε μια απάντηση η οποία βασίζεται σε στερεότυπα ότι όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν γίνει μέσα στην Αραβική Άνοιξη. Ξεχνάμε όμως συγχρόνως ότι όλες αυτές οι χώρες όπου υπήρξε η έκρηξη της Αραβικής ε, Άνοιξης. Έχουμε περάσει ήδη στο φθινόπωρο, ακόμα και στο χειμώνα. Όλες αυτές οι εξηγέρσεις έχουν περάσει αυτή τη φάση της άνθησης και είναι τώρα σε μια φάση κάμψης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορούσε να προβεί σε μια πιο επακριβή ανάλυση της κατάστασης στη Συρία. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές να μιλάει κανείς για τη βιαιότητα του καθεστώτος και να ζητάει την κατάλυση αυτού του καθεστώτος. Είναι πολύ πιο δύσκολο όμως να, κατανα... καταλάβουμε την φύση αυτής της κρίσης στη Συρία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι η Συρία είναι διαφορετική από τις άλλες χώρες του αραβικού κόσμου. Ήμουνα πρόσφατα με μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ισραήλ και άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση από ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ για τις ε, σχέσεις μεταξύ των ε, διαφόρων δογματικών ε, ομάδων. Είναι ένα μέλος της Κνεσέτ μάλιστα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν το οποίο θέλησε να μας δώσει στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ότι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να συμβεί μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Ασάτ. Πώς θα αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι μειονότητες, οι δύο σημειονότητες που υποστηρίζουν το, την τωρινή κυβέρνηση. Προφανώς ήξερα γιατί ομιλούσε <clears throat> και γιατί ανέφερε όλες αυτές τις ανησυχίες. Και φαίνεται ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επίτηδες έφερε ένα εκπρόσωπο του εκπρόσωπο του να μιλήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν είμαστε πάντα αρκετά αμερόληπτοι όταν μιλάμε για το, τη Συρία και τις διάφορες εξωτερικές επιρροές. Το Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία έχουν ένα συμφέρον στη Συρία και παίζουν και το παιχνίδι τους και μπορούν έτσι να επηρεάσουν ιδιαίτερα την κατάσταση. Μπορούμε να έχουμε ένα εμφύλιο πόλεμο, αλλά και ένα εμφύλιο θρησκευτικό πόλεμο μεταξύ Σουνιτών και Σιητών και υπάρξει και η προσπάθεια να περάσουν τα στρατηγικά συμφέροντα κάποιων μεγάλων δυνάμεων. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Όταν έχουμε την Κίνα και τη Ρωσία από τη μία πλευρά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι άδικο όταν εμείς αφήνουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα να τις πάρουν αυτοί, να τις δώσουν αυτοί οι οποίοι παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Η κατάσταση στη Συρία είναι όλο και χειρότερη. Δεν έχω αναφερθεί καν στην Αλκάιντα στη Συρία, στη δράση αυτής της οργάνωσης. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση λοιπόν η οποία επιτίθεται είναι η Αλκάιντα η οποία δεν επιτίθεται κυβέρνηση στον εαυτό της, είναι η Αλκάιντα που κάνει επιθέσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα αυτές τις πληροφορίες με ένα τρόπο ο οποίος είναι υπεύθυνο ως Ευρωπαίοι Κοινοβουλευτικοί και πρέπει να είμαστε τμήμα της παγκόσμιας πολιτικής. Εν τέλει, θα ήθελα να εκφράσω την αναγνώρισή μου, την ευγνωμοσύνη μου προς την Κομισιόν και την Γενική Διεύθυνση για τις ε, ανθρωπιστικές υποθέσεις και σε εσά κύριε Σόρενσεν προσωπικά γιατί έχετε με πολύ ευαίσθητο τρόπο μεταφέρει το μήνυμά σας σε σχέση με τις πολιτικές διαστάσεις αυτής της κρίσης και τον περιγύρο στον οποίο πρέπει να δουλεύετε. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς. Merci. Ευχαριστούμε ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσθέσει σε αυτό που ακούσαμε σήμερα αυτό. Ίσως η Κομισιόν απαντώντας να μας δώσει κάποια ένδειξη. Υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει και δεν έχει κάνει το Κοινοβούλιο για πόρους ή τέτοια, θα το καταλάβαινα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί και στην πρώην Ιουγκοσλαβία και το ρόλο που έπαιξε το ΝΑΤΟ κλπ. Για την επιβολή, όπως λένε, της ειρήνης. Νομίζω ότι η περιφέρεια ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε πάνω απ' όλα είναι να διατηρηθεί η εκεχηρία. Για ποιους λόγους ζητήθηκε η εκεχηρία. Τι έκαναν και οι δύο πλευρές. Υπήρξε και χειρία και δόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια ή όχι. Και περισσότερα, τι κάνετε για τις, με τις γειτονικές χώρες, η Ορδανία, Λίβανο, τους δώσαμε χρηματική βοήθεια, τους ρωτήσαμε ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς βλέπουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Κόρτες Λιστράδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Γιατί ο υπεύθυνο από την ΕΚΟ μας είπε να ανοίξει ο ανθρωπιστικός διάδρομος. Νομίζω ότι πολύ καλά το είπα, ότι πρέπει να υπάρξει αυτός ο προβληματισμός και συμφωνώ. Είναι μία προτεραιότητα να ανοίξει αυτός ο ανθρωπιστικό διάδρομος, αλλά πρέπει να υπάρξει απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που να έχει εγκριθεί από τη συνέλευση, από πλειοψηφία των χωρών εκεί. Μετά στο Συμβούλιο. Και αυτό έγινε. Στο Συμβούλιο όμως μετά η Κίνα και η Ρωσία μπλόκαραν την απόφαση. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ηθική υποχρέωση για μας να προχωρήσει αυτή η πρόταση. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κρίση στην Συρία. Και ίσως μάλιστα περισσότερο η Ρωσία από η Κίνα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Ίσως να είναι και η Ρωσία ένα στοιχείο κλειδί. Σας ρωτάω. Για να ανοίξει αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος. Πιστεύετε ότι όντω έτσι είναι. Στο τέλος, στο τέλος τέλος, είπατε και που μιλούσαμε για την Κίνα, Ρωσία και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, διακρίνοντας βέβαια την πολιτική από την ανθρωπιστική κρίση. Ε, λοιπόν, πείτε μας εσείς, πώς έχει αυτή η κατάσταση όταν μιλάμε για τη Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία. Τι δυνατότητες υπάρχουν να ανοίξει τελικά αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος που όλοι τον θέλουμε και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ανοίξει. Πρόεδρος, και εγώ έχω μία ερώτηση ή και δύο. 55.000 πρόσφυγες βλέπω στο έγγραφο ότι υπάρχουν στην Τουρκία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, ακόμα και στο Ιράκ. είναι μια ροή ανθρώπων πολύ φτωχών που δεν διαθέτουν καμία υποδομή, ούτε γεννήσει ούτε τίποτα. Και όταν βλέπω τις προσπάθειες που έγιναν για να βοηθηθούν, με εκπλήσει η μετριοπάθεια. Η Γαλλία 600 κουβέρτες έδωσε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω, η ΕΚΟ με τον ΟΙΕ φροντίζουν να υπάρξουν πραγματικοί καταφλισμοί με υπηρεσίες για αυτούς τους άτυχους ανθρώπους που μόλις ξέφυγαν από το θάνατο. Μπορούμε να τους προσφέρουμε υπηρεσίες υγιεινής, εκπαίδευση για τα παιδιά τους. Ποιος είναι υπεύθυνο για τέτοιους κατευλισμούς και εμεί η δικιά μας η Επιτροπή θα μπορούσε να επισκεφθεί τους πρόσφυγες αυτούς εκεί όπου βρίσκονται. Παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ε, ευχαριστώ για όλους σας για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και απαντήσεις που δεν τις έχω, γιατί δεν υπάρχουν βασικά. Καταλαβαίνετε ότι Μιλάω για την ανθρωπιστική πτυχή, όχι γιατί δεν μ' αρέσει η πολιτική, αλλά γιατί πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι προς το συμφέρον μου επίτηδες. Θέλω να κρατήσω διακριτές τις δύο δράσεις, την πολιτική και την ανθρωπιστική. Προφανώς το ειδευτικό σχέδιο του Κόφι Ανάν προέβλεπε έξι σημεία. Είναι μια πολιτική έτσι, η απόφαση. Το τέταρτο σημείο ήταν το ανθρωπιστικό, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει, αποτελώ μέρος της πρότασης αυτής. Και η ανθρωπιστική κοινότητα, όχι μόνο εμείς, αλλά και ο Ερυθρός Σταυρός κλπ. Έχουμε στηρίξει την προσέγγιση αυτή του Κόφιανάν. Η δουλειά του, εξάλλου, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες αλλά για να μιλήσουμε και λίγο για πολιτική, γιατί με ρωτήσατε. Η εκεχηρία ισχύει, δεν ισχύει. Μα βλέπουμε τι γίνεται επί τόπου. Δεν ισχύει. Ίσως, όμως, ίσως να υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη γιατί οι παρατηρητές του ΟΗΕ είναι στο δρόμο. Ενισχύονται. Αν λοιπόν ξεκινάνε από έξι... εννοείται δεν υπάρχουν ε, πολλές πιθανότητες. Αν όμως γίνουν 300, και τα νούμερα που έχω εδώ δείχνουν ότι έχουμε μια αύξηση. Άρα υπάρχει μια μικρή ελπίδα, έχοντας παρατηρητές επιτόπου, κάτι να γίνει με αυτή την εκεχηρία. Αναφέρεστε στους Κινέζους και τους Ρώσους. Εγώ μπορεί να έχω κάποια άποψη για την στάση τους στο Συμβούλιο Ασφάλειας, αλλά όσον αφορά την ανθρωπιστική πτυχή, ίσως μάλιστα ακριβώς επειδή κράτησαν τη στάση που κράτησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στην ανθρωπιστική πτυχή ήταν πιο βολική και μάλιστα ζήτησαν να βοηθήσουν περνώντας μηνύματα στον Ασάντα, στην κυβέρνησή του κλπ. Και δεν είναι τυχαίο που μετά από κάποιες συνομιλίες που είχαμε υπήρξε τελικά κάποιο άνοιγμα. Δεν είναι επειδή εγώ ο κύριος Όμερσον είπε κάτι, είναι επειδή το είπαν κάποιοι άλλοι που έχουν ε, πιο βαρύ λόγο. Νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε αυτό. Αλλά κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα για αυτά που λέτε για την πολιτική του στο σύνολό τη. Τώρα κύριε Ντεκάιζερ, ρωτήσατε και ζητήσατε διευκρινήσεις για το τι έγινε με τις διαπραγματεύσεις. Και μπορώ να σας πω ότι πράγματι Το θέμα είναι στο Ελίψ, τον Τάρα, στην Χόμς και στον Τάγια να έχουμε τέσσερα γραφεία. Και θα υπάρξουν άνθρωποι, όχι μόνο από εκεί, από την περιοχή, που να μην είναι ίσως εντελώς ανεξάρτητοι, αλλά θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν απ' έξω για να βοηθήσουν και να έχουν μια άποψη πιο ανεξάρτητη. Βλέπετε πώς γίνονται. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο η πόρτα αρχίζει να ανοίγει. Τώρα για τις γείτονες κυβερνήσεις. Και εδώ θα πω δύο λόγια. Είναι σαφές ότι οι πρέσβοι μας, οι επικεφαλής των ε, αντιπροσωπιών μας είναι σε συνεχή διάλογο με τις κυβερνήσεις της Λιβύης, της Ιορδανίας, της, της, της Τουρκίας. Με τις τρεις αυτές χώρες έχουμε προσφέρει μεγάλη βοήθεια. Για παράδειγμα στην κοιλάδα του Μπεκά, όπου δουλεύουμε με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχουν ε, πρόσφυγες, υπάρχουν ε, αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις εκεί, όπου κυρίως προσπαθούμε να βοηθήσουμε στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Ε, τα λεφτά προσπαθούμε να εκταμιεύονται ορθά. Και από εκεί και πέρα, αν μεθαύριο υπάρξουν και άλλα αιτήματα, εδώ είμαστε. Έχουμε σχεδιασμό. Στην Ιορδανία, επίσης, αυξήσαμε και εκεί τη στήριξή μας σε κάποιους καταβλισμούς. Στην Τουρκία είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί στην αρχή οι Τούρκοι φίλοι μας δεν θέλαν να πούν ότι υπάρχει στην επικράτειά τους ανθρωπιστική κρίση. Παρ' όλα αυτά βάλανε μπρο το Monitoring Information ε, System και έτσι βοήθησαν τέσσερις χώρες μέλη. Η Αυστριακή, αν δεν απατώμε, έστειλαν ένα κινητό νοσοκομείο, οι Γάλλοι, τα Ιταλοί. Πήγανε δηλαδή τα κράτη-μέλη και η Τουρκία είναι ευγνώμων. Αν μας ζητήσουν ανθρωπιστική βοήθεια, είμαστε έτοιμοι να την προσφέρουμε. Η κατάσταση στη Λιβύη, όπως είπατε, είναι πράγματι ιδιαίτερα περίπλοκη. Ό,τι κάνουμε εκεί είναι ότι δουλεύουμε με μέτρο. Δεν πρέπει να ορμήξουμε λέγοντας υπάρχουν πολλά προβλήματα, ε, διενέξεις, γιατί φυσικά και υπάρχουν με την κυβέρνηση, την Εσβολά κτλ. Αλλά πρέπει εκείνοι να έρθουν. Α, Λίβανο, έκανα λάθος, είπα Λιβύη, λέει ο μιλητής, έκανα λάθος, Λίβανο εννοούσα. Εννοείται ότι τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Και μας έρχονται εκθέσεις οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι εάν πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, θα έρθουν να μας το ζητήσουν. Κατόπιν τούτων, και επανέρχομαι στο πολιτικό σκέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολιτικό όργανο, οπότε δεν αρκεί να μιλάμε για το ανθρωπιστικό, πρέπει να μιλάμε και για το πολιτικό σκέλος. Αλλά ίσως δεν είμαι εγώ ο πιο κατάλληλος για να σας δώσω τέτοιες πληροφορίες. Χωρίς, και την άλλη μεριά σημαίνει ότι δεν θα βοηθούσα κιόλα αν έμπαινα πολύ στο πολιτικό σκέλος. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μας ε, βλέπουν απ' έξω ως ουδέτερους. Και πρέπει πραγματικά να μένουμε ουδέτεροι σε τέτοιου είδους σειράξεις. Ο κύριος Βάγκελ είχε πει ότι υπάρχουν πολλοί που παρεμβαίνουν στην κρίση αυτή. Είναι αλήθεια ότι αυτά που συνέβησαν πρόσφατα δεν είναι πράγματα απλά, αλλά εγώ, μια που ασχολούμαι με τα ανθρωπιστικά, δεν θα σχολιάσω από αυτόν. Αυτά είχα να σας πω. Καλή Merci beaucoup, Monsieur Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σόρενσεν.